Bueno, vamos a ir empezando. Καλησπέρα σα. Α αρχίσουμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε την απογευματινή δημόσια κρόση που θέμα έχει τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τα μέλη του πάνελ που θα μας διαφωτίσει σε ένα θέμα που είναι ύψης της σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η, Ευρωπαϊκή, η έχει πολλές διασυνδέσεις ε, και σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτοί που καταπολεμούν και αποκαλύπτουν τη διαφθορά, οι whistleblowers, αυτοί που καταγγέλουν απάτη ή διαφθορά, χρήζουν ιδιαίτερη προστασία. Αλλιώ είναι αδύνατο να πατάξουμε ουσιαστικά και στη ρίζα τη διαφθορά. Επίσης υπάρχει στενό σχετισμό. Ε, μεταξύ της διαφθοράς και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες. Οι ρίζες και των δύο φαινομένων είναι κοινέ. και σε μερικές περιπτώσεις η διαφθορά συνιστά καταστρατήγηση ειδικών δικαιωμάτων του πολίτη. Όλα αυτά θα τα πραγματευτούμε σήμερα, θα δούμε τις τάσεις που υπάρχουν, τις επιστάμενες προκλήσεις, το έργο που γίνεται από διάφορους φορείς, από διάφορε οργανώσει όπως τα Ηνωμένα Έθνη και θα εξετάσουμε και την εμπειρία συγκεκριμένων χωρών ή περιφερειών όπως είναι η κατάσταση στην Αφρική, η κατάσταση στη Γουατεμάλα, στην Ουκρανία ή στο Αζερμπαϊτζάν. Το 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σήμερα ε, βρισκόμαστε στη φάση επεξεργασίας της νέας έκθεσης για το θέμα αυτό η συγητής μας είναι ο κύριος Πέτρας Αουστρεβίτσιους, οπότε πριν να σας παρουσιάσω τα μέλη του πάνελ, του εμπειρογνώμονες μας, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αουστρεβίτσιους για να μας κάνει κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Madam Chair, colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που είναι πολύ βαθιά ριζωμένο ε, και μέσα αλλά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τον δείκτη της διαφθοράς ε, του 2015 δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στον κόσμο όπου να μην υπάρχει διαφθορά. Και δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την οικονομική ε, και πολιτική ανάπτυξη του κόσμου. Ε, οι κανονισμοί για την φοροαποφυγή, η εξαγορά ψήφων, ο χρηματισμός ε, στην οργάνωση αθλητικών ε, γεγονότων, αλλά και οι επιπτώσεις γενικότερα της διαφθοράς, όλα αυτά είναι λίγο πολύ τα ίδια. Όλα αυτά πάντα έχουν ένα τίμημα. Υπάρχει κατάχρηση εξουσίας για ε, προσωπικό όφελος και εις βάρος των υπολείπων, εις βάρος του ευρύτερου κοινού. Η διαφθορά λοιπόν εμφυλοχωρεί σε όλες ε, τις εκφάνσεις της ζωής ε, και προκαλεί ανισότητα και αδικία. Επηρεάζει τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και προς τους θεσμούς του κράτους και βεβαίως και προς το κράτος δικαίου. Έχει λοιπόν υπολογιστεί ότι η διαφθορά κοστίζει στον ε, ενωσιακό προπολογισμό μέχρι 990 δις, δηλαδή περίπου 1,3 τρεις ε, στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο. Ε, μπορείτε να καταλάβετε το τι συμβαίνει στον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο. Γνωρίζουμε ότι ε, το μητρό της διαφθοράς δεν λαμβάνει υπόψη του ότι υπάρχουν πολλές πρακτικές διαφθοράς ανά τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για να παρεμποδίσει και να προλάβει την διαφθορά. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά ε, κενά, παρατηράκια όπως λέγονται, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα όλων των ε, μέτρων κατά της διαφθοράς και να κρίνουμε κατά πόσον πράγματι είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά ή όχι και να κρίνουμε με βάση αυτά τα μέτρα την κοινωνία των πολιτών και γενικότερα την οικονομία με βάση πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Ε, το να είναι κανείς σε ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ε, το να είναι ενημερωμένη κοινωνία των πολιτών, αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη διαφθορά. Και ελπίζω στην έκθεση να αντιμετωπιστούν τα κενά. Προσβλέπω στο να συνεργαστώ με εσά και με τους συναδέλφους μου για να επιτύχουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και έχουμε ε, μία πολύ καλή ευκαιρία όχι μόνο να βελτιώσουμε την έκθεση του 2013 αλλά και για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και σε πολλούς άλλους τομείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα μας προσφέρεται η δυνατότητα να καλωσορίσουμε στο πάνελ μας ε, τους διακεκριμένους αυτούς αμπειρογνώμονες. Ε, πιστεύω ότι η προσέγγιση από το πριν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί διαφθορά και για να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά και προσβλέπω στο να ακούσω από εσάς ε, πολλές και διαφορετικές αναλύσεις ε, προσβλέπω στο να βελτιωθεί, να επεκταθεί περαιτέρω η έκθεση την οποία θα καταρτήσουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Οστρεβιτσούς. Η πρώτη μας ε, καλεσμένη είναι η καθηγήτρια Άννε Πέτερς που θα μας εξηγήσει το συσχετισμό της διαφθοράς με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μας παρουσιάσει τις νομικές πτυχές του θέματος και θα μας περιγράψει το έργο και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τα Ηνωμένα Έθνη στο τομέα αυτό. Η κυρία Πίτερς, η καθηγήτρια Πίτερς, είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Max Plan ε, για το Δημόσιο Συγκριτικό Δίκαιο και το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο και καθηγήτρια σε πολλά κορυφαία πανεπιστήμια και επικεφαλής πολλών ερευνών με το αντικείμενο αυτό. Κυρία Πίτερς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Είναι γνωστό, όπως αναφέρθηκε και από τον εισηγητή, ότι υπάρχει μια πραγματική σύμπτωση, ίσως και σχετισμό, γιατί οι χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς είναι αυτές που έχουν και τις πιο ε, χαμηλές επιδόσεις ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Αφγανιστάν, η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία είναι οι χαμηλότερε ε, σε ό,τι αφορά την αντίληψη ε, τη διαφθορά με βάση του δείκτε τη διεθνού ε, ε, διαφάνεια και έχουν προβλήματα με τη διαφάνεια και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φαίνεται ότι και η διαφθορά και η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευδοκιμούν στο ίδιο περιβάλλον και ίσω έχουν και τα ίδια αίτια, όπω είναι η φτώχεια και οι ασθενεί θεσμοί και οι καταστροφικές συνέπειες ε, της διαφθοράς, την ανάπτυξη, την εξάλληψη της φτώχειας, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια ε, δραστήρια πολιτική καταπολέμηση της διαφθοράς. Ε, έχουμε πολλές συμβάσεις σχετικές και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά εκθέσεις καταπολέμησης της ε, απάτης, της διαφθοράς και επίσης ε, υπάρχει το σχέδιο απόφασης, το πλαίσιο απόφασης για τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια, εδώ έχουμε περισσότερο το θέματα των, των, το τρίτων χωρών που αφορά περισσότερο όχι τόσο διαφθορά ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως δωροδοκία ε, από εταιρείε ε, με έδρα της Ηνωμένες, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση που λαμβάνουν μίζες, λάδωμα, φακελάκια κλπ δημοσίων υπαλλήλων σε τρίτες χώρες. Επίσης, έχουμε την σύμβαση του ΟΣΑ κατά της αλλοδαπής δωροδοκίας του 1997 και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση τη διαφθορά του 2003. Και μάλιστα η σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών είναι ανοιχτή στην πρόσβαση και για τοπικέ οικονομικέ οργανώσει, Από ό,τι ξέρω όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη συζητήσει την κύρωση τη σχετική σύμβαση του, όσα, του των Ηνωμένων Εθνών συγγνώμη, ως νομικό πρόσωπο. Και μάλιστα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2013 που ήδη αναφέρθηκε, αναφέρει το εξής. Η διαφθορά διαιωνίζει και επιδεινώνει αδικίες, ανισότητες και διακρίσεις ό,τι αφορά την, απόλαυση την ισότιμη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αναφέρει στο ψήφισμά σας του 2013. Και ακριβώς αυτή η γνώμη, δηλαδή ότι η διαφθορά, αν μη τι άλλο, επιδεινώνει τις παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι κοινή και σε άλλους ε, διεθνείς φορείς και οργανώσεις. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση της διαφθοράς που στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι στιγμής ε, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει δώσει εντολή στην Συμβουλευτική Επιτροπή για να διερευνήσει τον αρνητικό αντίκτυπο τη διαφθορά ό,τι αφορά την απόλευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα η τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκδόθηκε το 2015. Επίσης ζητήθηκε μια έκθεση για τις ε, βέλτιστες πρακτικές για να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα της διαφθοράς στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρεται μετά από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν μόνο 27 χώρε ε, κάποια αποτελέσματα. Βέβαια, Στι 27 αυτέ χώρε συμμετέχουν και κάποιες ε, σημαντικές για τον τομέα αυτό χώρε, όπως είναι η Ρωσική Ομοσπονδία και το Μαρόκο. Και μάλιστα οι κυβερνητικέ ε, δηλώσει συνοψίστηκαν και περιληφθήκαν στην έκθεση του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο και ανακεφαλαιώνει τις βέλτιστες πρακτικές. Τώρα, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη ε, προωθούν ε, αυτή την προσέγγιση που εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την προσέγγιση της διαφθοράς που εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί οι ειδικέ συμβάσει ε, για την καταπολέμηση τη διαφθορά είχαν μέχρι στιγμή απο χλωμά και απογοητευτικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι όλες οι συμβάσει που έχουμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που είναι 10-15, όχι μόνο οικουμενικέ αλλά και περιφερειακές, η περιοχή τη Λατινική Αμερική. παρόλα αυτά, παρά τι διεθνείς συμβάσει, ε, η διαφθορά σε μεγάλο βαθμό παραμένει ατιμόρυτη. Οπότε, εξού και η ιδέα της ανάγκης μιας νέας προσέγγισης. Όπως είπα, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι η διαφθορά ε, επιδεινώνει τη διάκριση σε ό,τι αφορά την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε διαρωτόμαστε, από νομική άποψη, η διαφθορά, οι διεφθαρμένες δράσεις ε, μήπως όχι απλώς επιδεινώνουν την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά παραβιάζουν συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κάποια κοινωνικά δικαιώματα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήδη η διαφθορά καταστρατηγεί τέτοια ειδικά δικαιώματα. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό το θέμα γιατί το να δείξουμε ότι η διαφθορά παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα ίσως δημιουργήσει ένα νέο σημείο εισόδου για, για τα εργαλεία και τα μέσα εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων για τη διαφθορά. Και έτσι γεφυρωθεί αυτό το γνωστό κενό της εφαρμογής ό,τι αφορά τις συμβάσεις κατά πολέμηση της διαφθορά. Ε, δύο ερωτήματα προκύπτουν εδώ. Το πρώτο είναι κατά πόσο μπορεί η διαφθορά να συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο ερώτημα που ε, είναι σημαντικό να το ε, επεξεργαστούμε είναι αν θα έπρεπε να ταξινομηθεί η διαφθορά ως ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό από κανονιστική άποψη το απάντημα στα ερωτήματα αυτά. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του πρίσματος της διαφθοράς στην κρατούσα πρακτική στα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιείται ένα πιο ήπιο, μια πιο ήπια ορολογία ε, για, το σχετισμό διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σχεδόν όλα τα κείμενα αναφέρονται στον αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα τα κείμενα αναφέρουν ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά από νομική σκοπιά είναι σημαντικό το κατά πόσο ε, χαρακτηρίζουμε μια κατάσταση ως ε, απλώς υπονομεύουσα τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αν θα τη χαρακτηρίσουμε ως ουσιαστική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε μπορεί να εμπίπτει στη χρήση των γνωστών μέσων και κυρώσεων που ισχύουν για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί συμπεριφορά ε, κρατική μιλάμε και να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών περιστάσεων. Έχουμε καταρχήν τη συγκεκριμένη διεφθαρμένη συμπεριφορά, το χρηματισμό αξιωματούχου που αποδίδεται στο κράτος, γιατί ο υπάλληλο αυτός, ο αξιωματούχο αυτός είναι δημόσιο υπάλληλο και δρά με δημόσια εξουσία. Το δεύτερο σημείο εισόδου είναι η γενική πολιτική πάταξη τη διαφθορά ε, τη χώρα ε, του κράτου ε, γενικώ και του κράτου ω νομικού προσώπου διεθνώ. Η ελληπής εφαρμογή μέτρων πάταξης διαφθοράς, ε, όπως αναφέρονται στη Διεθνή Σύμβαση, ε, συνιστούν παράληψη εκ μέρους του κράτους. Επίσης, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα προβλέπουν υποχρέωση του, της χώρας να δραστηριοποιηθεί. Οπότε η παράληψη της το συγκεκριμένο μέτρο, ίσω και αυτή συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, αποτελεσματικά μέτρα πάταξη διαφθορά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ω τρόπο για να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη με την υποχρέωση προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπω ξέρετε, όλα τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση ε, να προστατεύσουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα απέναντι σε τρίτους, ε, κυρίως οικονομικούς τελεστές. Και ε, ε, οικονομικούς ε, τελεστές που ε, επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά η υποχρέωση προστασίας απαιτεί από το κράτος όχι μόνο να προστατεύσει τους πολίτες από δράσεις άλλων ιδιωτών, όπως είναι κάποιοι οικονομικοί τελεστές, αλλά και να μειώσουν τους κινδύνους, τους διαφορετικούς κινδύνους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους οποίους συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι του κράτους αυτού σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιώματα που επηρεάζονται κυρίω από τη διαφθορά, για παράδειγμα το δικαίωμα στην υγεία, στην υγειονομική ε, περίθαλψη, το δικαίωμα στην παιδεία. Ε, το Διεθνέ Σύμφωνο για Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα περιλαμβάνει το άρθρο 2 και ένα γενικό κανόνα που αναφέρει ότι τα κράτη υποχρεούνται να εφαρμόσουν σταδιακά τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και επίση θα έλεγα ότι οι ορισμένε προποθέσει η διαφθορά και η ανοχή της διαφθοράς συνιστά καταστρατήγηση αυτής της υποχρέωσης ε, να εφαρμόσει προοδευτικά ε, μια χώρα τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ε, σε ό,τι αφορά την Διεθνή Επιτροπή για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη βασική υποχρέωση να λάβουν κάποια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα με σκοπό τη σταδιακή πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο συγκεκριμένο σύμφωνο, το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Οπότε τα μέτρα αυτά που περιλαμβάνει το σύμφωνο θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την άρση των εμποδίων για την υλοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων. Και η διαφθορά συνιστά τέτοιο εμπόδιο. Και ακριβώ επειδή συνιστά τέτοιο εμπόδιο, ε, θα πρέπει με βάση το σύμφωνο τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν μέτρα πάταξη τη διαφθορά. Η υπεξαίρεση, η κατάχρηση δημοσίων κονδυλίων, για παράδειγμα, σε υψηλό επίπεδο, παραβιάζει αυτή την υποχρέωση του κράτου. Γιατί σε τέτοιε περιπτώσει η χρηματοδότηση του βιωτικού επίπεδου υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων εμ, φαίνεται ότι υπερτερεί έναντι τη υλοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Άλλο σημαντικό θεωρητικό πρόβλημα για να, για να στοιχειοθετήσουμε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το θέμα της αιτιόδους συνάφειας. Θα πρέπει να αποδείξουμε αιτιόδη συνάφεια ε, της διαφθοράς με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι ε, μία από τις νέες αρχές ε, του νόμου για την κρατική ευθύνη είναι κάτι που θεωρείται εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση ή αναγκαιότητα και θα πρέπει να συμπληρωθεί από ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε ε, να κόψει τις αλυσίδες της αιτιόδου συνάφειας σε περίπτωση που είναι ειδικά ε, παρατεταμένες, μακριές Γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της ε, διαφθοράς αφενός και των αποτελεσματικών ή των ε, προβληματικών οικονομικών ή μορφωτικών υγειονομικών συστημάτων αφενός. Πώς θα αποδείξουμε λοιπόν την αιτιώδη συνάφεια. Θα πρέπει να, αποτελέσουμε, να αποδείξουμε ότι οι δεφθαρμένες δράσεις είναι εκ των όνων κανένα αλλά υπάρχει και μια εγκύτητα σε σχέση μεταξύ της ε, νομική παράβαση και της ε, παρεμπόδιση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, η άρνηση χορήγησης ιατρικού ραντεβού ή ενός πτυχίου από νομική άποψη συνιστά παραβίαση ανθρωπίνου δικαιώματος μόνο εφόσον η παράβαση αυτή είναι προβλέψιμη, σημαντικός αυτός όρος και όχι πολύ απομακρυσμένη από τη συγκεκριμένη δράση του διεφθαρμένου δημοσίου επαλλήλου. Για παράδειγμα, ε, φακελάκια που δίνονται σε ε, έναν υπάλληλο μιας ε, εποπτικής περιβαλλοντικής αρχής που στόχο έχουν να κάνουν τον υπάλληλο να παραβλέψει την ε, δημιουργία ενός παρα, μιας παράνομης χωματέρης τοξικών αποβλήτων με βάση τις αρχές αυτές αποτελεί αιτία των διαδοχικών επιζήμιων αποτελεσμάτων που έχει ενέργεια αυτή για τους κατοίκους της περιοχής. Δηλαδή, η διεφερμένη ανοχή του υπαλλήλου αυτού είναι για τον νόμο αιτία της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων της περιοχής ε, και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της ε, ε, σωματικής σωκεραιότητας. Το νέο θεωρητικό πρόβλημα είναι πού αποδίδουμε τη διεφθαρμένη συμπεριφορά, πώς αποδίδουμε τη διεφθαρμένη συμπεριφορά από τον υπάλληλο στο κράτος. Θα ήθελα τώρα να θέσω ένα ζήτημα για τη συζήτηση. Τη μορφή που ακούγεται πολλές φορές ότι μια τέτοια προσέγγιση που εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα πρόγραμμα της δύση και επιβολή των δυτικών αξιών και αρχών. Αυτή είναι μια επίκριση που ακούγεται για την προσέγγιση που εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιστική, αλλά θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη όταν μιλούμε για μια προσέγγιση της διαφθοράς που εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία καθηγητά. Δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αντουάν Τζιπλεσής που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου για την ασφάλεια στην Αφρική ε, μέτρα την Πρετόρια. Ο εμπειρογνώμονας μας έχει πολύ βαθιές γνώσεις ε, του φαινομένου της διαφθοράς στην Αφρική και την συνάρτησή της με τη δρομοκρατία καθώς και τις νέες απειλές στην ανθρώπινη ασφάλεια. Ο καθηγητής Ντυπλεσής ε, επίσης είναι επικεφαλής του τμήματος ε, για τις ε, διασυνοριακές απειλές και το διεθνές έγκλημα. Και για πάνω από μια εικοσαετία εργάστηκε σε θέματα ανθρώπινης ασφάλειας, καταπολέμησης του διεθνούς εγκλήματος και πρόθεσης δικαιοσύνης. Σε μια κοσαριά περίπου Αφρικανικέ χώρε, κορυφαίο εμπειρογνώμονα με βαθύτατες γνώσεις, ήταν και σύμβουλο των Ηνωμένων Εθνών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και με χαρά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντιπλεσής. Thank you very much. <clears throat> Truly is an honor to be... Ευχαριστώ και είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για κάτι που ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Άρχισα ως εισαγγελέα στην καριέρα μου πριν από λίγα χρόνια για το οργανωμένο έγκλημα. Δεν ήταν αυτός ο αρχικός στόχος, μηχανικός ήθελα να γίνω και μετά άκουσα τον Έλσον Μαντέλα να ε, μιλάει για τη σημασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποφάσισα να αλλάξω ε, και στην Νότια Αφρική δεκαετία των 90 να γίνει εισαγγελία. Ε, μετά το Απαρτχάιντ υπήρχε ένα κύμα ενθουσιασμού στη χώρα μας ε, σε σχέση με το τι μπορεί να σημαίνει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα για, την, ε, για το κοινωνικό σύμφωνο και για τη δημοκρατία. Ε, σε πάνω από 20 χώρες στην Αφρική έχω δουλέψει έκτοτε με διάφορες ιδιότητες με το ISS ή με τον ΟΗΕ ή με, ως σύμβουλος για κυβερνήσεις. Και το 2003 όταν συμμετείχα σε μια πολύ σημαντική περίπτωση διαφθοράς, δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε τότε τις ειδήσει, θα συνειδητοποιήσατε ότι πρόκειται για τα υψηλότατα κλιμάκια εξουσίας της χώρας μας και τότε είδα από κοντά πώς ε, συγκρούεται το δίκαιο με την εξουσία και συχνά πέφτει θύμα το δίκαιο. Ε, ε, τότε, εκείνη τη στιγμή, ή έκτοτε, να το πω καλύτερα, στη Νότια Αφρική καταφέραμε να δρομολογήσουμε και πάλι τη διαδικασία προς το κράτος δικαίου και όχι μόνο στη Νότια Αφρική αλλά και σε άλλες χώρες και ο ενθουσιασμός που έχω για αυτό το εργαστήρι και η, τον, νομική δυναμική του, της ενιολογικής, νέας ενιολογικής προσέγγισης της διαφθοράς μας ανοίγουν μια νέα στρατηγική, προοπτική στο, στρατηγική σημασία προοπτική στο, ζήτημα. Γιατί ασχολούμαι με το κράτος δικαίω διότι είμαι από αυτούς που εξακολουθούν να διαπνέονται από ενθουσιασμό για το μέλλον. Παρότι είναι πολλές και περίπλοκες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αφρικανική Ήπειρο ε, είναι πραγματικά ουσιαστικά τα προβλήματα, όμως στον πυρήνα πολλών προκλήσεων, είτε μιλάμε για συγκρούσεις, αγκαταγκαστική ε, μετανάστευση, ε, κλιματικές αλλαγές, στον πυρήνα βρίσκεται η διαφθορά και πολλοί εξακολουθούν να ε, θεωρούν ότι είναι ε, ε, η τάξη πραγμάτων, ότι έτσι ήθιστε να, να λειτουργούν όλοι στην Αφρική. Και μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη μάστιγα, ο μεγαλύτερος φωνιάς στην Αφρική είναι η διαφθορά και αν δεν αλλάξουμε κάτι θα συνεχίσει να ταλανίζει την Ήπειρό μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για τη σημασία του να επανεστιάσουμε την προσέγγιση δεν θα πρέπει να ακολουθούμε μόνο ε, την ε, ε, διάσταση της ποινική αντιμετώπισης διαφθοράς, αλλά να, όχι μόνο για ηθικούς λόγους, αλλά και για λόγους καλής στρατηγικής, επειδή υπάρχουν οι νέες επιταγές για όλες τις χώρες, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαχείριση παράνομης μετανάστευσης, επαγίωση της προόδου στην πορεία του εκδομακριτισμού. Και είτε μιλάω προς το εκπροσώπους του ιδιωτικού είτε σε εσά Μπορώ να σας πω ότι αυτή είναι η βέλτιστη προσέγγιση γιατί αν θέλουμε βιωσιμότητα ε, και ειρήνη ε, σε οποιαδήποτε χώρο, οποιαδήποτε ήπειρο θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Νομίζω ότι είναι προοδευτικός ο τρόπος ε, που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις και φυσικά είναι η διαφθορά άνευ προηγούμενη αποδεκατίζει το δικαστικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή. Όμως αντιστέκονται και αντιμάχονται αυτό το φαινόμενο οι Νοτιοαφρικανοί και ε, το συνταγματικό μας δικαστήριο είπε χαρακτηριστικά σε μια πολύ σημαντική υπόθεση όπου εμπλέκεται και ο πρόεδρος μας, είπε το εξής. Δεν μπορεί να υπάρξει κέρδος αν η διαφθορά απειλεί οτιδήποτε μας είναι αγαπητό, οτιδήποτε αν απειλεί τη συνταγματική τάξη, το, τη δημοκρατία, ε, τις βασικές δημοκρατικές αρχές, στο κράτος δικαίου και τις αξίες ε, της συνταγματικής πορείας της χώρας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι η απάτη, οι παραβάσεις, η ολιγορία, από πλευράς του κράτους δεν επιτρέπουν να εφαρμόσουμε τις ε, συνταγματικές αρχές της χώρας μας. Είναι πολύ προοδευτική αυτή η δήλωση και όχι μόνο επειδή έρχεται από την ανώτατη δικαστική αρχή, αλλά από πλευράς πολιτικής, από πλευρά αντίδραση όπως ακούσαμε και για το συνταγματικό δικαστήριο της Ινδίας νομίζω ότι υιοθετεί μια ε, σύγκρισιμη προσέγγιση. Η διαφορά δεν είναι μόνο αφρικανικό είναι ή νοτιοαφρικανικό το πρόβλημα, δεν θα πρέπει να το πιστέψει κανείς. Ε, σίγουρα δεν είναι, αλλά ε, λειτουργεί ω καταλητική δύναμη για την τρομοκρατία για άλλα προβλήματα όπως η μαζική ε, μετανάστευση ή ε, τα προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε να γράψουμε τη συζήτηση σε ένα διαφορετικό πλαίσιο ούτως ώστε πέρα από τους νομικούς μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τις ευκαιρίες ε, ούτως ώστε η κοινωνία των πολιτών να έχει στην διάθεσή της τα απαιτούμενα μέσα για την αντιμετώπιση διαφθοράς. Ε, και νομίζω ότι είναι πολλοί που δεν εννοούν να το καταλάβουν, να καταλάβουν αυτή την αλλαγή, ε, ότι έχει τα τελευταία χρόνια ε, αποδοθεί αυξημένη έμφαση στην ε, καταπολέμηση της διαφθοράς και υπάρχουν μέσα που μέχρι στιγμής χρησιμοποιούσαμε τα οποία δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και αν εξακολουθήσουμε με αυτή την αμυγό ποινική προσέγγιση δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα εξακολουθούν να υποφέρουν ε, τα θύματα της διαφθοράς και φυσικά στην καρδιά του προβλήματος είναι ε, και η πολιτική βούληση, τα συμφέροντα ε, και διαπλεκόμενα συμφέροντα κυβέρνηση και ιδιωτικού τομέα είναι στην καρδιά του προβλήματος. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που συναντιούνται ε, η εξουσία και το δίκαιο. Και νομίζω ότι η προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική αρχή. Βλέπουμε ότι εφαρμόζονται οι αρχές από τις εμβάσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, σε παγκόσμιο επίπεδο, περιφερειακές οργανώσεις, ε, το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας, ε, παραδείγματος χάρη, ε, ο ΙΕ, έχουν τις συμβάσεις που θεσμοθετούν το πρόβλημα, την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά δεν διαθέτουν κυρώσεις λοιπόν. Ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν διάφορα είδη ευθύνη σε σχέση με τα ανθρωπινά δικαιώματα που αγγίζουν τα κράτη τα ίδια, τις κυβερνήσεις των κρατών, όπως σωστά είπε το Συνταγματικό Δικαστήριο. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μηχανισμό για να ανταποκριθούμε. Αν δούμε τώρα την Διεθνή Σύμβαση, ε, βασίζεται στη συνένεση και ε, για να εφαρμοστεί πρέπει να δράσουν τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει αποτελεσματικέ κυρώσει σε περίπτωση παραβίαση τη σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα φόβο δίωξη ή επιβολή κυρώσεων. Η πολιτική βουλήση λοιπόν δεν επαρκεί στα πλαίσια αυτή τη προσέγγιση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Ε, υπάρχουν πολλά που μπορώ να πω και δεν ε, εννοώ ότι πρέπει να ε, καταργήσουμε την προσέγγιση ε, των ποινικά κολάσιμων πράξεων και τη ποινική ψυχική εδίωξη, αλλά θα πρέπει να, ή την εστίαση για την κατάσχεση, τη δίμευση, τον επαναπατρισμό των προϊόντων ε, παρανομών δραστηριότητων. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν. Φυσικά στα πλαίσια τη ποινική δικαιοσύνη, θα πρέπει να αυξήσουμε τα ένδικα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν αρκεί όμω αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη δίωξη και στη, ε, από την εισαγγελία ε, των διαπλεκομένων. Θα πρέπει τα, από τη, στην κοινωνία των πολιτών οι υπερασπιστές καταπολέμησης αυτού κινούμε Οργανισμός τη διαφθορά να μπορέσουν να έχουν μέσα στη διάθεσή του, να υποχρεώσουν τι κυβερνήσει, ούτω ώστε να πληρούν τι του τους υποχρεώσεις ε, ε, και έτσι να καταπολεμήσουν τις, καλύτερες, τις μεγα, κάποιου κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για αυτή την προσέγγιση που εστιάζεται γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να το επαναλάβουμε ότι χρειαζόμαστε μέσα. Ε, προτού περάσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, παρότι υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση κινούνται σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν συγκλίνουν οι πορείες αυτές οι δύο προσεγγίσεις παρόλα αυτά εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο δηλαδή την καταπολέμηση διαφθοράς λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, θα πρέπει με κριτικό πνεύμα να εντοπίσουμε τα πεδία που μπορούμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας, ε, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες, ε, τα δίκτυα που έχουν οι μεν και οι δε για την εκπληρώση του ίδιου στόχου. Για να κάνω συγκεκριμένες συστάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε, τουλάχιστον ε, στην Αφρική, να, το διάλογο και να ευθυγραμμίσουμε το διάλογο να, για να μπορέσουμε να περάσουμε σε πράξεις και υπάρχουν σε νομικό, θεωρητικό, ε, ιδεολογικό και ε, ε, πολιτικό πεδίο διάφορα επιχειρήματα, διάφοροι τρόποι για να εντείνουμε τη συνεργασία μας, να αναπτύξουμε νέα προγράμματα, να έχουμε κοινή χρηματοδότηση σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε πολυμερές ε, ως προς το διάλογο για τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα προγράμματα που μπορούν να εφαρμόσουν ε, θα, επίσης. Ε, επειδή προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει ο ΙΕ το ζήτημα ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον ΙΕ και να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία είναι και τα δίκτυα, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει εξ αρχής τη δέσμευση με βασικούς εταιρούς από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχουν τρία βασικά στρατηγική σημασία ζητήματα για την Αφρική, Αφρικανική Ένωση, γιατί αυτή είναι η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιούμε, αλλά φυσικά και στη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς, όπως σας είπα. Είναι πολιτικά ε, φορτισμένο αυτό το ζήτημα, ε, παρά το νομικό χαρακτήρα του και αναγνωρίζοντας και το ρόλο του ιδιωτικού τομέα, όπως σωστά είπατε και στην παρουσίασή σας. Επίσης, ε, νομίζω ότι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρειαζόμαστε πρωτόκολλα τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν σε όλα τα προγράμματα αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να δίνεται αυτή η εντολή σε όλε τι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην Αλοδαπή. Τέλο, για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, Χρειάζεται σταδιακά να δράσουμε, ε, διότι πρόκειται για ριζική αλλαγή, τη ε, ε, αλλαγή της προσέγγισης που επιδιώκουμε. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και από τη ρίζα προς τα πάνω θα, με συζητήσεις, με φόρα, διάλογο, να εμπλακούν οι άνθρωποι, να σου αποδείξουμε ότι λειτουργεί αυτή η νέα προσέγγιση για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με, την, με τα παραδοσιακά δίκτυα. Και ε, μπορούμε να ε, επιδιώξουμε ένα νέο ανθρώπινο που δεν θα έχει αυτή την τάση, την έμφυτη τάση για τη διαφθορά. Και επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη ε, στο εσωτερικό των χωρών τους ε, να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους με συγκεκριμένες δράσεις, ούτως ώστε για αυτή την παγκόσμια βιλή να μπορούν να συγκλίνουν με άλλες χώρες που ενστερνίζονται τις ίδιες ιδέες και να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα σε μια σύνδεση μέσω Skype με τον κύριο Μανφρέντο Μαροκίν Βοχόρκεθ που είναι πρόεδρος ε, της δράσης των πολιτών, ο τοπικός εκπρόσωπος ε, της Διεθνούς Διαφάνειας στη Γουατεμάλα. Δυστυχώς η σύνδεση δεν είναι και πολύ καλή. Η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά, αλλά χωρίς διερμηνία. Γιατί είναι πολύ ε, κακός ο ήχος μέσω Skype για διερμηνία.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 Σας συγχαίρω θερμότατα για το έργο σας, πραγματικά αξιέπαινο σε μια χώρα με αρκετά δύσκολη κατάσταση. Πάντως δείξατε την ε, αδειάστη δέσμευσή σας ε, υπέρ της, υπέρ της πάταξης της Τώρα αλλάζουμε ήπειρο τελείω και θα ακούσουμε τον κύριο Ίγκορ Τσερνιάκ που είναι αντιπρόεδρος της μη κυβερνητική οργάνωσης κέντρο καταπολέμησης της διαφθοράς ε, της πόλης Χάρκοβο στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, Όλες οι χώρες μας ενδιαφέρουν εννοείται. Αλλά ακριβώ επειδή είναι η των χώρα με σημαντική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή για την πρόθεση των απαραίτητων αλλά δύσκολων μεταρρυθμίσεων που καλείται να πραγματοποιήσει, και επίσης εμπλεκόμαστε και στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο κύριος Τσένεκ θα μας παρουσιάσει την κατάσταση στην Ουκρανία και θα μας δώσει και ε, μια τοπική προοπτική της πατρίδας, της γενέτειρας του Χάρκοβο, στην οποία εκλέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 2015. Κύριε Τσέρνικ, σας ακούμε. Uh, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, αγαπητοί μετέχοντες, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που μου προσφέρετε η ευκαιρία για να σας ενημερώσω για τον αγώνα κατά της ε, διαφθοράς στην Ουκρανία. Η διαφθορά θεωρώ ότι είναι από τα βασικότερα προβλήματα στην Ουκρανία. Στον Ιούνιο έγινε μια έρευνα και τα στοιχεία που προέκυψαν είναι χαρακτηριστικά. Το 39% των Ουκρανών θεωρούν ότι το υψηλό επίπεδο διαφθοράς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ουκρανίας και η επιθετικότητα στην Ντομπάς απασχολεί βέβαια τους Ουκρανούς περισσότερο από την Ουκρανία. Στην Ουκρανία υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διαφθορά τα τελευταία 20 χρόνια και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, επεκτάθηκε η στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία και αυτό αποδεικνύει ότι ισχύουν, ε, ισχύει το άρθρο 8 ε, του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό το λόγο το να υπάρχουν ουσιαστικέ μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, αυτό είναι το βασικό καθήκον των οργανών της Ουκρανίας. Όμως οι αρχές της Ουκρανίας ε, κατανοούν πολύ καλά πως θα πρέπει να να εκπλώσουν τις δικές τους τις υποχρεώσεις. Και μερικές φορές μοιάζει απλά να μιμούνται, να προσποιούνται ότι αγωνίζονται κατά της διαφθοράς. Ε, παράδειγμα, ε, η εφαρμογή ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος για την υποβολή δηλώσεων στην Ουκρανία. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος είναι προαπαιτούμενο για να πάρει κανείς ε, οικονομική βοήθεια από από τους εταίρους της Ουκρανίας. Ο νόμος σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2014 προβλέπει ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα ε, που θα ξεκινήσει το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, στις 18 Δεκεμβρίου του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια θετική έκθεση σχετικά με το πώς εφαρμόζει η Ουκρανία το πρόγραμμα δράση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Το πιο σημαντικό έλαβε όμως χώρα στις 25 ε, Δεκεμβρίου του 2015 ε, στο κοινοβούλιο μας θεσπίστηκε μία τροπολογία η οποία καθυστερεί την ε, εφαρμογή του συστήματος του ηλεκτρονικού μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. Βεβαίως οι αντιδράσεις της ε, κοινωνίας στην Ουκρανία και των εταίρων ήταν πάρα πολύ αρνητικοί. Έτσι λοιπόν το Μάρτιο του 2016 οι αρμόδιες αρχές ε, αναγκάστηκαν να κυρώσουν αυτή την τροπολογία και φαίνόταν ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εφαρμογή του νέου συστήματος, αλλά αυτά δεν συμβαίνουν στην Ουκρανία. Είχε προβλεφθεί ότι το σύστημα θα εγκατασταθεί στις 15 Αυγούστου, αλλά στις 2 Αυγούστου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα κυρίως σε έναν δημόσιο φορέα ε, στο να χορηγεί ε, ένα πιστοποιητικό. Ο αγώνας λοιπόν για αυτό το πιστοποιητικό συνεχίστηκε για κάποιες εβδομάδες. Ε, δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να λυθεί το πρόβλημα. Από τις 15 Αυγούστου αυτό το ε, πιστοποιητικό δεν υποβάλλεται. Στην πρακτική εφαρμογή αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν είναι αρμόδιος ε, σχετικά με την ε, ακρίβεια της του συστήματος. Έτσι λοιπόν ο νόμος για την πρόληψη της διαφθοράς ε, έγινε πλέον ε, ανυπόστατος. Ε, το θέμα είναι ότι δεν μπόρεσε να εγκατασταθεί το σύστημα στις 15 Αυγούστου. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις και την ίδια ακριβώς ημέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Οι αρχές Ουκρανίας υποσχέθηκαν να θα βρουν μια γρήγορη λύση. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Είναι αύριο, η 1η Σεπτεμβρίου, άρα δηλαδή σε λίγες μόνο ώρες θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι αρχέ τη Ουκρανία εκπληρώνουν τι υποχρεώσει του ή όχι. Η κατάσταση όσον αφορά αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα αντιλώσεων είναι ο κανόνα και όχι η εξαίρεση. το ηλεκτρονικο συστημα δηλώσεων άλλο παράδειγμα είναι μια κατάσταση που προέκυψε πρόσφατα σε σχέση με το γραφείο κατά τη διαφθορά στην Ουκρανία. Αυτό το γραφείο είναι ένα φορέα που έχει συσταθεί για να εξετάζει ε, περιπτώσει διαφθορά. Και λόγω τη θέση των Ευρωπαίων εταίρων και του ρόλου πολλών ακτιβιστών, το γραφείο αυτό έχει συσταθεί με βάση τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς που αναφέρονται στο άρθρο 29 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γραφείο κατά της διαφθοράς ε, άρχισε την ποινική δίωξη κατά πολλών στελεχών, κυρίως του Κωνσταντίν Κουλίκ, που είναι ένας ε, από τους ε, στρατιωτικούς δικαστές στην Ουκρανία. Υπάρχουν υποψίες εναντίον του για εμπλουτισμό. Αυτός όμως δεν έδωσε καμία εξήγηση για το πού βρήκε όλα αυτά τα πολυτελή διαμερίσματα σε μια πολύ καλή περιοχή ε, και τα πολυτελή αυτοκίνητα που ανήκουν στην οικογένειά του. Και παρά τις ε, ε, αγωγές αυτός όμως παραμένει στη θέση του. Οι σχέσεις τώρα ανάμεσα στο γραφείο κατά διαφθοράς και του συγκεκριμένου τρόπου έφτασαν στο να εγκλειστούν στη φυλακή δύο, δύο υπάλληλοι, χαμηλότεροι υπάλληλοι και τους ασκήθηκε και σωματική βία για να αποκτηθούν στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αγώνας κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία σε γενικές γραμμές σημαίνει στεναρή αντίδραση της ε, παλιάς ε, διεφθαρμένης ε, ελίτ. Η κατάσταση στο Χάρκι είναι ακόμα πιο συγκεκριμένη. Τα τελευταία οκτώ χρόνια το Χαρκίβ βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο μιας πολιτικής ομάδας, ε, το οποίο βρίσκεται στον έλεγχο του ε, Γιόρκιτς. Ε, επίσης, ε, ο δήμαρχος έχει εκλεγεί από το 2010, ο Χέναντι ο οποίος είναι συνώνυμο της διαφθοράς για πάρα πολλούς. Ε, σήμερα ε, συνδέεται το όνομά του και με, το, με την αντίσταση ο κύριος Κέρνες εξακολουθεί να έχει την πλήρη εξουσία. Ε, το, η δουλειά του Κέντρου κατά της διαφθοράς και μια δική μου οργάνωση που εκπροσωπώ έχουν ως στόχο να εκτέσουν τον Δήμαρχο και τα προγράμματά του κατά της διαφθοράς. Αυτό ενδιαφέρει είναι να προβάλλουμε τους μηχανισμούς καταχρήσεων στον προπολογισμό του Δήμου. Έχουμε κάνει πάρα πολλές έρευνες που αφορούν στην εταιρεία Parking Plus και χάρη των Panama Papers μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στους συνεταίρους του κυρίου Κέρνες και των ε, πρωθυπουργό της Ρωσίας, τον κύριο Μετβέντεφ. Αυτή η εταιρεία έχει λάβει 80 εκατομμύρια Αμερικάνων δολάρια από τον προπολογισμό του Δήμου τα τελευταία 8 χρόνια και επ' αυτού έχουμε καταθέσει αγωγές σε διάφορες αρμόδιες αρχές. Περιμένουμε τώρα το αποτέλεσμα των ερευνών. Το δικό μας το κέντρο επίσης έχει συμμετάσχει στην αποκάλυψη ενός άλλου μεγάλου ε, προβλήματος διαφθοράς που αφορά στις, σε χωροταξικά προβλήματα στο Χάρκοβο. Η περιοχή ε, η οποία μετατράπηκε παράνομα και μεταφέρθηκε παράνομα από το Δήμο σε εμπορικούς οργανισμούς ε, είναι πολύ μεγαλύτερη από 500 εκτάρια, δηλαδή ε, τέσσερις φορές το, του Μονακό, της έκτασης του Μονακό. Η ζημιά που προκλήθηκε είναι περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια και πρέπει να πω ότι δεν μας εξέπληξε όταν διαπιστώσαμε ότι οι βασικοί αποδέκτες έχουν άμεση σχέση με τον Δήμαρχο, τον Κέρνης. Ε, αυτή τη στιγμή ε, οργανισμοί αρμόδιοι ερευνούν την περίπτωση αλλά το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί και γι' αυτό το λόγο με την υποστήριξη του ε, Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία ξεκινήσαμε την αναθεώρηση των αποφάσεων του Δήμου σχετικά με την απαλωτρίωση αυτών των εκτάσεων. Ε, το δικαστικό σύστημα στην Ουκρανία καθιστά όμως σχεδόν αδύνατο για μία ΜΚΟ ε, να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ξεκινάμε τώρα μία εκστρατεία έτσι ώστε να στηρίξουμε τις νομοθετικές αλλαγές που θα επιτρέψουν σε μη κυβερνητικού οργανισμούς να έχουν εξουσία για τη δικαστική προστασία των πολιτών. Ε, οι έρευνε, οι δημοσιογραφικέ κυρίω είναι το βασικότερό μας εργαλείο για να προστατεύσουμε τους πολίτες, αυτούς που φύγονται από τη διαφθορά. Και έτσι λοιπόν κατορθώσαμε ως κέντρο να επιτύχουμε τη μία πώληση ενός υπαλλήλου ο οποίος ε, είχε κατηγορηθεί, την απόλυση μάλλον του υπαλλήλου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για διαφθορά. Το δικό μας το κέντρο ε, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και αυτό μας ανησυχεί. Από την άλλη πλευρά όμως ε, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και για να ανακεφαλαιώσω θα ήθελα να επισημάνω ότι μόνο η, ε, η συστηματική πίεση στις Ουκρανικές αρχές μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να προηγούνται και μόνο εφόσον είναι επιτυχημένες, μόνο τότε θα μπορεί κανείς να μιλάει για οικονομική βοήθεια. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή την αρχή που προκύπτει από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Υπάρχουν όμω τρία θέματα που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση στον αγώνα κατά τη διαφθορά και να προάγουν ουσιαστικέ αλλαγέ στη ζωή των ανθρώπων που υποφέρουν από τη διαφθορά. Το πρώτο είναι η νομιμοποίηση των ΜΚΟ, να μπορούν αυτέ να έχουν δικαστική αναθεώρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται. Δεύτερον, ε, να από ποινικέ ευθύνε εκείνοι οι οποίοι ε, βοηθούν στο να αποκαλύπτεται διαφθορά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιου είδου προβλέψει, ε, πρόνοιε ε, στην νομοθεσία τη Ουκρανία. Τρίτον, σαφή διάκριση των εξουσιών ανάμεσα σε φορεί που επιβάλλουν τον νόμο και στο σύστημα ελέγχου που έχει προκύψει από τη θέσπιση του νέου νόμου για ε, την εισαγγελία. Αυτά τα τρία μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα. Δεν πρόκειται μόνο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και για την ε, προστασία των πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσέρνιακ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρεμπέκα Βενσόν Δεν ξέρω, προφέρω, το προφέρω στα γαλλικά, Βενσά, αλλά μπορεί να είναι και Βίνσεντ. Η κυρία Ρεβέκα Βίνσεντ είναι συντονίστρια της Συμμαχίας Αθλητισμός για τα Δικαιώματα. Και μάλιστα ξεκίνησε εκστρατεία κατά της διαφθοράς και της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως στο Αζερβαϊτζάν. Όπως ξέρετε, στις μεγάλες αθλητικές ε, ε, ε, εκδηλώσεις έχει νόημα να κάνουμε μια ενδελεχή ανάλυση της δέσμευσής τους, της στράτευσής τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σχέση τους με τη διαφθορά. Πολλές φορές ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, της, ε, του συσχετισμού δηλαδή του αθλητισμού με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα θέλαμε να ακούσουμε την κυρία Ρεμπέκα Βινσέντ που θα μας παρουσιάσει το έργο της Συμμαχία Αθλητισμός για Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ευχαριστώ. Κύριε Βενσάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τη Red for Sport Coalition, συνασπισμό ε, διεθνών ε, ΜΚΟ μικρών ε, που συνεργάζονται για να επιστήσουν την προσοχή στι περιπτώσει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Αρχίσαμε ω ακτιβιστέ που διώκονταν ή φυλακίστηκαν στι χώρε του ή στο Μπακού στην Ελβετική Ψβία είχαν καταφύγει για προστασία. Έχει έρθει ο συνάδελφο μα να σα τα πει σήμερα και αρχίσαμε αυτή την καμπάνια για τη, τα ε, πρωταθλήματα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε πέρσι στο Μπακού και μιλάω για πολλές αθλητικές εκδηλώσεις όπου τίθεται τέτοια ζητήματα. 15 μήνες μετά δυστυχώς η κατάσταση μάλλον έχει χειροτερέψει. Το ε, στο Αζερμπαϊτζάν. Παραδείγματο χάρη για όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε για τη διαφορά και τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί αυτά τα δύο ζητήματα είναι αλληλένδετα και υπάρχουν σοβαρότατε περιπτώσει. Ε, υπάρχει σε συστημικό επίπεδο κάλυψη και ε, υποστήριξη ε, τέτοιων ε, διεφθαρμένων διαδικασιών και επίσης τον Grand Prix της Φόρμουλα 1. με την αθλητική αυτή εκδήλωση επιταχύνθηκε αυτό το φαινόμενο της διαφθόρα στο Αζερμπαϊτζάν. Το καλό είναι ότι η διεθνή κοινότητα, τα διεθνή ΜΜΕ έστρεψαν το βλέμμα τους σε αυτή τη χώρα και έτσι αναμετέδωσαν ειδήσει και μπόρεσαν, μπόρεσε και το ευρύτερο κοινό να γνωρίζει την κατάσταση Χρειαζόμαστε όμως συγκεκριμένη δράση, ώστε οι αρχές ε, του Αζερμπαϊτζάν να ε, καταστούν υπόλογες για τις πράξεις τους. Είναι από τις πιο διεφθαρμένες χώρες του κόσμου, ε, από την διεθνή διαφάνεια, από 168 χώρες βρίσκεται στην 119η θέση η θεση χωρα και από το Human Rights ή από τους Ρεπόρτες Χωρίς Σύνορα, που είναι και μέλη της οργάνωσής μας, είναι στην 163η ε, θέση από ε, τις 180 συνολικά για την ελευθερία τύπου. Πάνω από μία δεκαετία η ε, οικογένεια του Ελ Χαμαλή του Προέδρου και άλλοι διαπλεκόμενοι έχουν επεξαιρέσει δισεκατομμύρια από τη χώρα και ΜΜΕ όπως η Radio Free Europe, η Radio Liberty αναμεταδίδουν τέτοιες ε, ειδήσει. Ε, ξέρετε την Καντίζα Ισμαήλοβα, είναι μια γνωστή δημοσιογράφος, συνάδελφο που πλήρωσε βαρύτατο το τίμημα για το κουράγιο που είχε να ε, μεταφέρει τι ειδήσει για αυτό το ζήτημα στο Αζερμπαϊτζάν. Έγινε απόπειρα εκβιασμού. Το 2012 οι αζερικές αρχές ε, την ε, πίεζαν για πολλά χρόνια και το 2012 το Μάρτιο πήρε ένα φάκελο με προσωπικές της φωτογραφίες ε, που την απειλούσαν ότι θα τη διασύρουν αν δεν σταματήσει. Με θάρρος συνέχισε, εξέδεσε τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Αζερμπαϊτζάν και τελικά την συνέλαβαν το Δεκέμβρη του 2014 και μετά καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια κάθεριξη για οικονομικούς ε, λόγους, ε, κατηγορίες. Ή ε, πρόκειται για μηχανογραφία που κατασκεύασαν τις κατηγορίες και τελικά τον Ιούνιο του 2015 απελευθερώθηκε η Καντής. Είναι τυχερή από αυτή την άποψη γιατί δεν είναι στη φυλακή, δεν μπορεί να ταξιδέψει βεβαίως. Αυτό είναι σύνηθες. Πολλοί Αζέρι δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα για πολιτικούς λόγους. Η Καντίτσα λοιπόν ε, ε, είναι σε μια μεγάλη φυλακή σε ολόκληρο το Αζερβαϊτζάν. Μη θεωρείτε δηλαδή ότι το, με την απελευθέρωσή της βελτιώθηκε η κατάσταση. Όχι. Η Κατήτσα είναι από τις πιο προεξέχουσες φυσιογνωμίες που απελευθερώθηκαν ε, φέτος. Ε, υπάρχει εντύπωση ότι βελτιώθηκε η κατάσταση, ότι υπάρχει μια θετική τάση ε, και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι και τις τελευταίες εβδομάδες που ήμασταν όλοι διακοπές, οι αρχές συνέχισαν την καταστολή τους παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά που συμβαίνουν είναι συγκρίσιμα με τις εξελίξεις στην ε, Τουρκία. Ε, ε, ε, δημοσιογράφοι συνελήφθησαν διότι, στην Τουρκία έτσι για την, διότι συνδέθηκε το όνομά τους με τον Γκουλάν αλλά αυτό είναι μία πρόφαση μόνο ε, μια σκευωρία και στις 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει ένα δημοψήφισμα και πάλι θα σιγά, θα, ε, ε, με εκφοβισμό θα καταστήλουν οποιασδήποτε φωνές αντίστασης για, να κερδίσουν το δημοψήφισμα. Εκατοντάδες περιπτώσεις δημοσιογράφων κρατούνται στη φυλακή εδώ και χρόνια. Ίγμα Μαρ Κάντοφ είναι ο ηγέτης της Πολίτευση, εναλλακτικό δημοκρατικό κίνημα, μισή χρόνια στη φυλακή, δεν υπάρχει ε, ε, πολιτικά κατασκευασμένες κατηγορίες, ε, παρότι έχει εκδοθεί εντολή για την απελευθέρωσή του, κρατείται ακόμη. Η Νατίτσκα Φόλη πρόσφατα απελευθερώθηκε από το ίδιο κίνημα σε αυτό το νέο κύμα καταστολής και αντιμετωπίζει σοβαρότητα τις κατηγορίες. Ο Ζάρτη επίσης blogger, ακτιβιστής τρία χρόνια, ζέμαρχαζή, δημοσιογράφο, δημοσιογράφος που πριν από δύο χρόνια γιορτάζει την, δεύτερη, την, επέτειο, τη δεύτερη επέτειο για την σύλληψή του. Ε, Κιάζη Ιμπραχήμοβ, Αμάντοφ, Γκαραμόν. Ε, όλα αυτά είναι ονόματα των νέων πολιτικών κρατωμένων. Υπάρχουν και επίσης ε, ε για βασανιστήρια. Ε, Φαγή Κναμύροφ, άλλη μια περίπτωση, αντιμετωπίσω αντιμετωπίσει ε, απειλή για ε, πολιετή κάθριξη ε, και επίσης ε, μέσα που υποχρεώνονται να σταματήσουν την, τις εκδόσεις τους, έντυπες εκδόσεις τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κράτος προσπαθεί να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι τελείως ο κατάλογος και οποιαδήποτε αντίποση και αν έχουν κάποιοι ότι βελτιώνεται η κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν, λυπάμαι που θα πω, δεν ευσταθεί και θα πρέπει ε, να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της διαφθοράς ε, για να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Ε, υπάρχουν ναι, μεμονωμένες κυρώσει ε, κατά των αξιωματούχων που συμμετέχουν ε, σε αυτές τις παρεμβάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, σχετικό είναι και ένα πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι κατακρίθηκε από πολλούς αλλά από πλευρά διεθνή κοινότητα είναι το ισχυρότερο ψήφισμα που είδαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν και τα ονόματα των φίλων μου που ήταν μέσα στο ψήφισμα εκτιμούν την υποστήριξή σα μέσα από το ψήφισμα, καλωσορίζουν αυτή την ιδέα των προσωπικών κυρώσεων κατά ε, των ε, αξιωματούχων τη ε, κυβέρνηση και ζητούν να συνεχίσετε τι προσπάθειε σα. Οι μεμονωμένε ατομικέ κυρώσει νομίζω θα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση τη διαφθορά στο Αζερβαϊτζάν και το προτείνουμε και σε άλλα μέρη, όπω τι είπα, παραδείγματο χάρη, τη πράξη Μαγνίσκη ή το ψήφισμα για τη δημοκρατία στο Αζερβαϊτζάν. Όλα αυτά είναι εργαλεία που πιστεύουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ούτω ώστε να λογοδοτήσουν ε, στην, ε, στην Αμερική οι αξιωματούχοι ε, που έχουν εμπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις στο Αζερβαϊτζάν. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα για μεταρρυθμίσεις στο Αζερβαϊτζάν. Αυτή τη στιγμή συζητείται η Συμφωνία Πλαίσιο για το Αζερβαϊτζάν και θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία μέχρι ότου να εφαρμοστούν συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει, αρχίζοντα βέβαια από την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, κατάργηση επιθετική νομοθεσία, κατάργηση τη απαγόρευση ταξιδιού για εξέχουσε φυσιογνωμίε και τώρα είναι ε, σημείο καμπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δυνατότητα να ασκήσει πίεση στο Αζερβαϊτζάν. Η διεθνή κοινότητα χρειάζεται περισσότερο, λένε κάποιοι το Αζερβαϊτζάν, παρότι το αντίθετο. Αυτό δεν ισχύει. Αζερβαϊτζάν χρειάζεται και τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω τώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δράσουμε. Νομίζω εξέπνευσε ο χρόνο που μου αναλογούσε. Θα σταματήσω. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ. Και τελευταίο μα καλεσμένο. είναι ο, ο κύριος Κρίστοφ Κλέριξ που θα μας παρουσιάσει τη φωνή των δημοσιογράφων. Ο Κρίστοφ είναι δημοσιογράφος του περιοδικού ΚΝΑΚ, βελγικό περιοδικό. Ε, γνωρίζει τον κόσμο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και έχει πάρει και βραβείο από την ε, Φλαμανδική Ένωση Δημοσιογράφων το 2015 και θα μας παρουσιάσει, θα μας εξηγήσει τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αυτά που μάθαμε μετά τη Swiss Leaks και τα έγγραφα του Παναμά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλό σας απόγευμα. Είναι ιδιαίτερη χαρά για ένα δημοσιογράφο να μιλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εμεί ω Διεθνής Όμιλο Ερευνητική Δημοσιογραφία ε, βλέπουμε ότι αναγνωρίζετε το έργο, μου, το έργο μα ε, και πολύ σπάνια ε, έχουμε την ευκαιρία να φέρνουμε άρθρα στο Κοινοβούλιο για να τα συζητούν οι πολιτικοί. Εγώ λοιπόν εργάζομαι για το ΚΝΑΚ στο Βέλγιο, αλλά είμαι και μέλος τη Διεθνούς ένωση Ερευνητικής Δημοσιογραφίας ε, που συστήθηκε πριν από 20 χρόνια από τον Charles Lewis ε, και τώρα έχει γίνει και μία μικρή ε, μικιό με την έννοια ότι υπάρχουν 11 αμοιβόμενοι δημοσιογράφοι. Ε, ξεκινήσαμε με 76 δημοσιογράφους σε 41 χώρες ε, και εντωμεταξύ έχουμε 200 δημοσιογράφους από 65 χώρες. Ε, περίπου το 1 τρίτο των κρατών του κόσμου εκπροσωπούνται. Τώρα, τι συμβαίνει. Εγώ δουλεύω για το ΚΝΑΚ και όταν εμφανίζεται ένα θέμα που αφορά την ένωσή μας, με ενημερώνουν, ε, το ΚΝΑΚ εξακολουθεί να πληρώνει το μισθό μου, ε, το ΚΝΑΚ αποφασίζει ε, τις ιστορίες που θα δημοσιεύσουμε, βρίσκω πληροφορίες από τη Διεθνή Ένωση και συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου. Έτσι λοιπόν λειτουργεί το όλο θέμα. Πληρώνομαι από το περιοδικό μου, αλλά είμαι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ερευνητικής Δημοσιογραφίας. Τρία πράγματα είναι σημαντικά πριν ξεκινήσουμε ένα project. Εξετάζουμε θέματα που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο ε, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αν δει κανεί ε, τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι καταφέραμε να ξεκινήσουμε ε, με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διεθνές offshore companies, οι εξωχώριες εταιρείε, ε, περίπου 20.000 είναι εξωχώριες εταιρείε και οι πληροφορίες ήρθαν από δύο εταιρείε. Μία από τη Σιγκαπούρη και η άλλη από το BVI. Το επόμενο που ακολούθησε ήταν οι διαρροές του Λουξεμβούργου το 2014, πάλι φορολογία, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με εξωχώριες, αλλά με μυστικές φορολογικές συμφωνίες που συνήφθησαν ανάμεσα στις αρχές του Λουξεμβούργου και 300 εταιρείε από άλλα μέρη του κόσμου. Ε, οποίο ε, έγινε και μία πολύ σημαντική έρευνα ε, τα Swiss Leaks ε, το 2015 Φεβρουάριος αποκαλύφθηκαν περίπου 80.000 μυστικοί λογαριασμοί της HSBC στην Γενέβη και από εκεί 102 δις δολάρια εμφανίστηκαν. Και τέλος η τελευταία έρευνα που ακολούθησε μέχρι τώρα είναι τα Panama Papers, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο αυτού του έτους. 3 Απριλίου του 2016 βλέπουμε ε, εφημερίδες από ολόκληρο τον κόσμο που δημοσίευσαν τις ιστορίες για τις εξωχώρες εταιρείε και ήταν η μεγαλύτερη διαρροή πληροφοριών που συνέβη ποτέ. Άρα δηλαδή μιλάμε για ιστορική συνεργασία κάτω από αυτό το πρίσμα. Αν δείτε λιγάκι αυτή την εικόνα το βλέπετε. Cable Gate ήταν 1,7 gigabyte όταν δημοσιεύτηκαν από τα Wikileaks, offshore leaks, 260 gigabytes και τα Panama Papers ήταν τεράστιες πληροφορίες, 2,6 ε, terabytes και τα μισά εξ αυτών ήταν από email, τα άλλα από X-Files Μπορείτε να δείτε εδώ τα στοιχεία PDF, εικόνες και το καθεξής. Όλες αυτές ήταν πληροφορίες που αφορούν σε εξωχώριες εταιρείες. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα μέσα ενημέρωση που υπήρξε από 476 δημοσιογράφοι που εκπροσωπούσαν 109 μέσα ενημέρωση από 76 χώρε και η έρευνα διήρκησε ένα χρόνο. Δουλεύαμε μυστικά πριν ε, δημοσιεύσουμε τις ιστορίες μας από τον Απρίλιο και εντεύθεν. Βλέπετε λοιπόν και κάποια παραδείγματα των εγγράφων που διέρευσαν 11 εκατομμύρια, σαν παράδειγμα, Αυτά είναι αρχεία τα οποία διέρευσαν από τις ε, εταιρείε αφορούν σε εξωχώριες εταιρείε. Οι εξωχώριες εταιρείε είναι το βασικό μας θέμα. Και οι εμπειρογνώμονε μας λένε ότι υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πολύ συχνά ε, καταφεύγουν ε, σε νομοθεσίε με χαμηλή φορολογία και το δεύτερο είναι ότι οι εξωχώριες εταιρείε τώρα μπορούν να συστήνονται ανώνυμα. Εγώ είμαι Βέλγος δηλαδή, αν ε, πάω στο Βέλγιο να συστήσω μια εταιρεία, και υπάρχει κάποιο ίχνος δικό μου. Αλλά αν συστήσω εξωχώρια με κάποιες ε, νομοθετικέ διευκολύνσεις, μπορώ να το κάνω χωρί να αφήσω κανένα ίχνος πίσω μου ότι εγώ είμαι ε, ο αποδέκτης ε, και ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού που έχει σχέση με αυτή την εταιρεία. Άρα δηλαδή οι εξωχώριες παρακάμπτουν την νομοθεσία. Εγώ το είπε κάποιο πολύ απλά. Ποτέ δεν έχω δει κάποιον για να συστήσει μία εξωχώρια για να είναι διαφανής. Κάτι θέλει να κρύψει. Δεν σημαίνει ότι αυτό ε, γίνεται πάντα, ε, την παράνομο. Ας πούμε ότι κάποιος είναι πολύ πλούσιος και φοβάται τους εκβιασμού, θέλει να τα κρύψει. Ή κάποιοι που είναι σε διάσταση για τα διαζύγια, θέλουν να κρύψουν στοιχεία από τον ή τη σύζυγο. Αλλά συνήθως οι προθέσεις δεν είναι τόσο διαυγή. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι μια εξωχώρια δεν είναι παράνομη στο βαθμό που δηλώνει κανείς ε, τα κεφάλαια αυτής της εφόσον τη δηλώνει αυτήν και ακολουθεί και τους κανόνες του παιχνιδιού. Δουλεύει κανείς ε, με πραγματικούς υπαλλήλους, όχι με εταιρείε ε, εικονικές. Πρέπει όλα να είναι νόμιμα. Και όμως στην περίπτωση αυτή θα διερωτηθούμε, μα γιατί να τα κάνει κανείς όλα αυτά από τη στιγμή που έτσι κι ε, μπορεί να δηλώσει το κεφάλαιό του με πολύ πιο απλό και νόμιμο τρόπο. Όσον αφορά τη Μόσακα Φωσέκα ε, στον Παναμά, είναι μια νομική εταιρεία και γι' αυτό μιλάμε για Panama Papers, αλλά προφανώς ο Παναμάς δεν είναι η μόνη χώρα που επιτρέπει στην νομοθεσία του τους εξωχώριες. Όμως εδώ ε, η διαρροή έγινε από τον Παναμά, γι' αυτό μιλάμε για Panama Papers. Βλέπετε εδώ την ε, άνοδο και την πτώση της Μόσακ Φωσέκα. Ε, θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ πρόκειται για μία από τις βασικότερες ε, ε, εταιρείε που συστήνουν εξωχώρηση ανά τον κόσμο, αλλά δεν είναι μόνη. 11 εκατομμύρια έγγραφα διέρευσαν από αυτή την εταιρεία. Και από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στα Panama Papers, είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξωχωρίων. Και να το ξέρετε αυτό, γιατί εμείς ήδη δημοσιεύσαμε πάρα πολλές ιστορίες για πολιτικούς. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι το παγόβουνο. Αν εδώ μιλάμε μόνο για την κορυφή. Στην προηγούμενη ε, διαφάνεια βλέπετε ότι μιλάμε για 200.000 εταιρείες που συστήθηκαν με τη βοήθεια της ε, Μόσαχα Φωσέκα. Το 2010 ήταν η απόλυτη ε, αποκορύφωση και μετά σιγά σιγά υπάρχει μία μείωση. Το είπα λοιπόν ότι ο Παναμάς δεν είναι ο μόνος που επιτρέπει τέτοιου είδους νομοθεσία. BVI ε, στην περίπτωση αυτή μιλάμε για πάνω από 200.000 εταιρείε. Ακολουθεί μετά ο Παναμάς, μετά ακολουθούν ο Παναμά, ε, οι Σεχέλες και το καθεξής. Mossack Fonseca BVI. αυτό μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα αν αναζητήσετε εξωχώριες εταιρείε. Και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τις, ε, τα Panama Papers, όπως ε, σας είπα, ε, διέρευσαν περίπου 11,5 εκατομμύρια έγγραφα. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 14.000 εξωχώρες εταιρείε. Δεν είναι μόνο εταιρείε, είναι εταιρείε καταπιστεύματα και ιδρύματα. Βρήκαμε έγγραφα που διέρευσαν για αυτά τα τρία τρεις μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πάντως, αν θέλει κάποιος ε, να συστήσει μια εξωχώρα, θα πάει κατευθείαν στην ε, δικηγορική εταιρεία τη Φορσέκα, θα δουλέψει πρώτα ο ενδιάμεσος ε, που είναι ο ε, τραπεζίτης, ο δικηγόρος, αυτοί όλοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και έχουμε εντοπίσει 14.000 ενδιάμεσους οι οποίοι βοηθούν στη σύσταση των εξωχών εταιριών. Πάρα πολύ φορολογική παράδειση, ε, πάνω από 10. Εμείς ε, εντοπίσαμε 12 αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων, 60 συγγενείς τους, πάνω από 140 πολιτικούς και στελέχη αυτοί όλοι αποκαλούνται PAPs, Politically Exposed People. Οι τράπεζες ε, θα πρέπει λοιπόν να δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους PEPs και δεν είναι ε, πρόβλημα απαραίτητα το να έχει ένας πολιτικός μια ξεχώρια, αλλά το να έχει αυτομάτως δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Μέχρι τώρα έχουμε βρει 29 ε, δισεκατομμυρίουχος της, ε, του καταλόγου Forbes ε, που έχουν συστήσει εταιρείε στον Παναμά, έχουν σχέση με τα Panama Papers και για άλλη μια φορά θέλω να υπογραμμίσω το ρόλο των ενδιάμεσων. Εδώ υπάρχει μια ειδική κατηγορία. Μιλάμε για τράπεζες. Πάνω από 500 τράπεζες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία διότι ε, είναι ενδιάμεση, όπως σας είπα, ανάμεσα στη ε, δικηγορική εταιρεία και τον τελικό πελάτη. Ανακαλύψαμε πάνω από 50.000 εξωχώρες εταιρείες, οι οποίες έχουν συστηθεί από τράπεζες και ενδιάμεσους. Και βλέπετε κάποιες εικόνες εδώ των πολιτικών που ενεπλάκησαν ε, θα έχετε όλοι ακούσει μάλλον ε, την ιστορία του ε, Πρωθυπουργού της Ισλανδίας, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί λίγες μόνο μέρες μετά τις πρώτες δημοσιεύσεις, ο Κουν Λάξον και ο κυρίως επίσης Πέτρο Ποροσέγκο, Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, πρόεδρος μάλλον της Ουκρανίας, Μπορείτε μόνοι σας να τα δείτε λιγάκι αυτά και να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις ιστορίες με όλες τις λεπτομέρειες. Κατόπιν, αν δούμε τον ρόλο των τραπεζών, σας είπα ότι πάνω από 500 τράπεζες εμπλέκονται. Εδώ βλέπετε τις 10 ε, σημαντικότητες. Αν δείτε την πρώτη, η Εξπέρτα, είναι μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο που έχει ε, βοηθήσει να συσταθούν πάνω από 1.600 εξωχώριες εταιρείες. Η Εξπέρτα τότε ήταν υποκατάστημα ε, ενός βελγικού τραπεζικού ομίλου. Η Εξπέρτα είναι και μια κοινοβουλευτική επιτροπή, έτσι λέγεται, εξετάζει τα Panama Papers και οργανώνει και ακροάσεις. Ε, το καλό, η καλή είδηση είναι ότι κάποιες από αυτές τις πληροφορίες δημοσιεύτηκαν. Ε, εμείς αποφασίσαμε αυτά τα 11 εκατομμύρια έγγραφα, να μην τα ε, δημοσιεύσουμε όλα και αυτό για διάφορους λόγους, γιατί υπάρχουν και θέματα ε, ιδιωτικής σφαίρας, αλλά από την άλλη η Διεθνής μας Ένωση έχει ε, δημοσιεύσει τις βασικές πληροφορίες για τις εταιρείες που εμπλέκονται. Βασικές πληροφορίες σημαίνει ότι αυτά που θα τα έβρισκε κανείς ε, ε, στο κανονικό μητρό ε, μιας χώρας, ποιος είναι δηλαδή ο πρόεδρος, ποιος είναι ο γενικός διευθυντής μιας εταιρείας, όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεθνούς μας Ένωσης και έτσι οι φορολογικές αρχές μπόρεσαν να ξεκινήσουν τις έρευνες. Αν δείτε μετά τις επιπτώσεις των Panama Papers που δημοσιεύτηκαν πριν από τέσσερις περίπου μήνες, ε, θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για το Ρεκιαβίκ, τη Μάλτα και το Λονδίνο. Χιλιάδες ανθρώπων ε, κατέβηκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν και ως αποτέλεσμα αυτού ε, παρετήθηκε ο Πρωθυπουργό της Ισλανδίας, στην Ισπανία παρετήθηκε ένας υπουργό, έγιναν απολύσεις στην Ολλανδία, ε, στην Αρμενία παρετήθηκε ένας ε, στρατηγός, στην FIFA ένας, ένα μέλος της, Επιτροπής, της Διοντολογικής Επιτροπής. Ο Ντέβιτ Κάμερον ανακοίνωσε ότι θα λάβει νέα μέτρα για τη διαφάνεια. Οι φορολογικές αρχές των περισσότερων χωρών ήρθαν σε επαφή μαζί μας από το Βέλγιο αλλά και πολλές άλλες χώρες που αναφέρονται εδώ στο κατάλογο τις βλέπετε τις χώρες αυτές στη διαφάνεια. Η δική μας η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα πρωτότυπα έγγραφα αλλά πολλές σημαντικές πληροφορίες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας. Εκτός από τις φορολογικές έρευνες που ξεκίνησαν, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες έρευνες που δρομολογήθηκαν σε άλλες χώρες ε, Παραδείγματο χάρη ε, για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Συστήθηκαν κοινοβουλευτικές επιτροπές, έγιναν ε, έρευνες σε πολλές χώρες, Αργεντινή, Δανία και σε πολλές άλλες χώρες. Ελβετία, στην Ουρουγουάη συνελήφθησαν πέντε άτομα ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά. Βλέπουμε ότι πολλοί είχαν έρθει σε επαφή με το οργανωμένο έγκλημα και ε, διαπιστώθηκε ότι από τη στιγμή που είναι κανείς διατεθειμένος να κάνει μία σοβαρή ποινική έρευνα, κατά κανόνα καταλήγει σε εξωχώριες εταιρείε. Και αυτό είναι δύσκολο και για τους εισαγγελείς, για τους ε, ποινικά εμπλεκόμενους ε, γιατί χρειάζονται πάρα πολλές ειδικέ γνώσεις. Ε, υπάρχουν εξωχώρες εταιρείε ε, οι οποίες ευημερούν. Θεωρώ λοιπόν ότι το κλειδί αυτής της ομιλίας πρέπει να το έχετε κατά νου είναι ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι η λύση του προβλήματος. Σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα επιτρέπονται ίσως πλέον οι εξωχώριες εταιρείε, αλλά μέχρι να ζήσουμε αυτό τον αγγελικά πλασμένο κόσμο ε, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Ε, Παραδείγματο χάρη, βελγικέ φορολογικέ αρχέ ή ε, οι ανακριτέ να μπορούν να απευθυνθούν απευθεία στον Παναμά. Και στην περίπτωση αυτή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι πληροφορίε για εξωχώριε εταιρείε θα στέλνονται απευθεία στο Βέλγιο. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι όλη η ιδέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει ε, μια επιτροπή, θα ξεκινήσει αργότερα, στο τέλος του μήνα, θα ερευνήσει τα Panama Papers. Νομίζω λοιπόν ότι αν δει κανεί ε, το αποτέλεσμα, σε τέσσερις μήνες έχουν γίνει πάρα πολλά. Εμείς ε, προσβλέπουμε και σε άλλα αποτελέσματα από τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει ολόκληρο το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ναγκόμες, που είναι η προηγούμενη συγκήτρια της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που οργανώσατε αυτή τη δημόσια κρόση υπό την αιγύδα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ευχαριστώ τους καλεσμένους για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, και αλληλοσυμπληρούμενες παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπε ο κύριος Κλέριξ. Το θέμα αυτό σκόταν ήδη στο επίκεντρο της πρώτης έκθεσης ε, για το σχετισμό διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς από το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί όπως είδαμε από τα στοιχεία που μας δώσατε και από τις αποκαλύψεις που έγιναν από τα έγγραφα του Παναμά και τις σχετικές διαρροές, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και υπάρχουν πολλά στρώματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της διοχέτευσης των αυτοκοδηλίων, της τροφοδότηση διαφθοράς και της ε, καταστρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η πρώτη μεγάλη τράπεζα του Λονδίνου που εμπλέκεται εξυπηρετούσε ακόμη και την βασιλική οικογένεια. Επίσης και η Deutsche Bank έχει αφιερώσει 10 δισεκατομμύρια για να βοηθήσει κάποιες ε, μυστικές υπηρεσίες να, να συστήσουν εξωχώριες. Δεν είναι θέμα μόνο πίεση. Θα πρέπει να το ελέγξουμε το δικό μας τραπεζικό σύστημα και το δικό μας λογιστικό σύστημα, το σύστημα λογιστών, δικηγόρων, ε, οικονομικών συμβούλων. Είναι όλοι κεντρικοί παράγοντες, πρωταγωνιστές ε, σε αυτούς τους, ε, σε αυτούς τους διάβλους της διαφοράς που έχουν ταυτόχρονα επιζήμιες συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τους whistleblowers, ε, τους θαραλέους αυτούς καταγγέλλοντες από τη Γουατεμάλα που καταπολεμούν την ατιμορρησία, τους ανθρώπους από το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία που κάνουν ό,τι μπορούν, που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Και η περίπτωση της Ουκρανίας είναι ενδεικτική θα πρέπει να βρίσκεται συνέχεια στο επίκεντρο της προσοχής μας και πολλά χρήματα που έχουν επεξεραθεί από το προηγούμενο καθεστώς και έχουν κλαπεί από τους φορολογούμενους περνάνε μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάμειξη των ευρωπαϊκών φορέων των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, των Ευρωπαίων Δικηγόρων και ακόμη χειρότερα είναι το θέμα με την Ουκρανία γιατί ο Πόρτνοφ ε, ουσιαστικά μας κοροϊδεύουν, μας περιγελούν, μας πιάνουν κορόιδο γιατί έχουν καταφέρει να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες εις βάρος τους. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί στις ε, έρευνές μας στην Εξεταστική Επιτροπή και θα το κάνουμε επ' ευκαιρία τον εγγράφο του Παραμά. Επίσης σήμερα παρακολουθήσαμε την περίπτωση της Apple, της Apple που θα αναγκαστεί να πληρώσει ε, φόρους επιτέλους γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε για μια φορά αυτό που όφιλε να κάνει γιατί αυτό θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καθήκον της να αναλάβει δράσεις και αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό χάρη στις αποκαλύψεις που έγιναν από τα LuxLeaks και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκθέσεις το, δύο εκθέσεις των Επιτροπών Τάξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι ασκήσαμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζητήσαμε εντόνως να αναλάβει δράση και να στηρίξουμε την Επίτροπο στο έργο της. Χάρη στη, στα LuxLeaks και το έργο της Επιτροπής φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για την υποχρέωση της Apple να καταβάλει φόρο στην Ιρλανδία. Επίσης, ε, θα πρέπει ε, ο συσχετισμός διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής μας και να τονιστεί δεόντως. Επίση, αναφέρθηκε το θέμα του, ξέπλυμα, του ξεπλήματος χρήματος, ε, νομοποίησης εισόδων από παράνομε δραστηριότητε και τη ανάγκης ε, τη δέουσα επιμέλεια εκ μέρου του τραπεζικού συστήματο. Υπάρχει μια διεστραμμένη συνεργασία εδώ που επιτρέπει αυτές οι εικονικές εταιρείε ή τις εταιρείε γραμματοκιβώτιο ε, που έχουν μείνει στα ράφια για πολλά χρόνια να αναφέρουν απλώς ένα διευθυντή που κρύβει ουσιαστικά πολλούς πίσω του. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε ε, ποιος είναι διευθυντής, είναι το θέμα ποιοι βρίσκονται πίσω από το διευθυντή. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες αυτών των ε, εταιριών και πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Κύπρος, ε, όλες σχεδόν έχουν αυτό το διαστραμμένο σύστημα το φορολογικό ώστε να επιτρέπουν το απόρριτο ε, της κυκλοφορίας αυτών των χρημάτων. Επίσης, μιλούμε για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όχι μόνο εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτές οι παραβιάσεις που γίνονται στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες ε, γιατί αυτά τα μέτρα λιτότητα έχουν στερήσει ανθρώπινα δικαιώματα από πολλού. έχουν στερήσει πρόσβαση στι υπηρεσίες υγεία, στην παιδεία και υπάρχουν αυτά τα μέτρα και αυτή η καταστρατήγηση γιατί ακριβώ δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα στα φορολογικά συστήματα γιατί είχαν διαρρεύσει προς φορολογικού παραδείσους. Μιλάμε λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πάταξη τη διαφθορά και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ναι, δεν είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και το φαινόμενο, αλλά είμαι σχεδόν βεβαία ότι πολλά χρήματα από το Αζερβαϊτζάν, από τη Γουατεμάλα, την Ουκρανία ή την Αγγόλα στην ουσία έχουν ξεπληθεί μέσω των ευρωπαϊκών τραπεζών, επενδύονται στις επιχειρήσεις και στα οικοπεδά μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπα ισχύει αυτό στην περίπτωση της Πορτογαλίας και ασχολούμαι ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και η διαφθορά και όσοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η της διαφθοράς και οι υπέτειοι της παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ελέγχουν τις τράπεζες και ουσιαστικά ε, λιμένονται την κατάσταση και συνεχίζουν αυτή την συμπεριφορά την εγκληματική. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε δράση είναι καθήκον μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτος είναι ο κύριος Ρικάρδο Σέρβι, ματάρχης του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολυμερούς Διπλωματίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια εγώ και μετά θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμπληρώσει την παρουσίαση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την οργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης, γιατί όπως ε, συμβαίνει πολύ συχνά ε, στις συζητήσεις ε, στην Επιτροπή σας για συγκεκριμένα θέματα, είναι τόσο ευρεία και ευρυθής η προσέγγιση που γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και για μας. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η νέα προσέγγιση, το νέο σημείο εισόδου για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, του σχετισμού διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτή την συνάφεια, της, το σχετισμό μεταξύ διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι σχετικά κάτι καινούργιο και για μας, γιατί όπως σας είπα ε, προερχόμαστε από διαφορετικές κοινότητες και ε, αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Τα επισήμανε και η κυρία Αναγκόμε το ζήτημα είναι τεράστιο και οριζόντιο και είναι πολύ δύσκολο μερικέ φορές να επικεντρωνόμαστε σε ένα και μόνο θέμα και να έχουμε καλό συντονισμό. Είναι δύσκολο να βρούμε κάποιον από την ΕΕΔ που θα καλύπτει όλες τις πτυχέ αυτού του πολυσχεδούς ε, φαινομένου. Πάντως, εγώ εξετάζω το θέμα υπό τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η οπτική γωνία και είναι σημαντικό που αυτό το πρίσμα χρησιμοποίησαμε στη σημερινή συζήτηση. Και έχουμε και εμείς την ευκαιρία να διδαχθούμε πολλά πράγματα με μια τόσο εκτενή παρουσίαση των εμπειριών και συγκεκριμένων χωρών για το, τη σχέση διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως, ε, εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε κυρίως, ε, να διδαχθούμε, να μάθουμε, να ακούσουμε και τις νέες προσεγγίσεις που προτείνονται. Και σε ό,τι αφορά την γενικότερη πολιτική που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2015-2019, σχετικά καινούριο, μόλις τώρα γιόρτασε την πρώτη επέτειό του και καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων και προτεραιοτήτων αυτό το σχέδιο δράση για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το βασικό έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδυάζει ουσιαστικά τι προσπάθειε όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Και από τι βασικέ προτεραιότητε στο σχετικά καινούριο αυτό ε, σχέδιο δράση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι επικεντρώνεται στην ενίσχυση των τοπικών θεσμών, των ε, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και φυσικά την ενίσχυση της ε, στήριξης των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο ε, του σχεδίου δράσης, αλλά υπάρχει κάποιο περιθώριο να περιλάβουμε και τις δραστηριότητες πάταξης της διαφθοράς. Γιατί είναι σημαντικό το σχέδιο δράσης να προωθεί τη σύσταση ειδικευμένων φορέων ε, που θα καταπολεμούν ε, τοπικά τη διαφθορά. Θα ακούσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι συγκεκριμένες μας δράσεις σε επιμέρους χώρες Πάντω, έχουμε ω γενική προτεραιότητα του σχεδίου δράση για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα την ενίσχυση τη εμπειρογνωσία ε, και τη ικανότητα ε, των τοπικών φορέων να πατάξουν τη διαφθορά αναπτύσσοντα πολιτικέ χρηστή ε, διαχείριση των δημοσίων πόρων. Αυτό είναι μία από τι βασικέ μα προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ΤΕΦΟ, κυρία Αλεξάνδρα Μιάτσα. Uh, Ευχαριστώ και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον ε, συγητή και τους διακεκριμένους προσκεκλημένους. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και των προκλήσεων αλλά και συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι γιατί ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση, οπότε μάλλον είναι και σωστή. Εξυπακούεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στον πυρήνα της ε, αναπτυξιακή συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε εταίρου. Καθηγητή Πίτερ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που κάνατε. Η διαφθορά είναι μέγιστη τροχοπέδη για την υλοποίηση των σχεδίων μας για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πολιτιστικά, κοινωνικά, ε, ε, ε, κοινωνικά δικαιώματα και ταυτόχρονα να επιτύχουν ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες. βασικές αρχές όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η απουσία διακριτικής μεταχείρισης και ταυτόχρονα ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά είναι εργαλεία ε, πολύ σημαντικά στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Για να καταπολεμήσουμε λοιπόν αποτελεσματικά τη διαφθορά, χρειαζόμαστε αποτελεσματικά θεσμικά όργανα, ε, καλή νομοθεσία κρατικές μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα συμμετοχή όλων των φορέων, κυβερνητικών και μη. Υποστηρίζονται οι δράσεις κατά τη διαφθοράς, όπως είπε ο συνάδελφος, σε διάφορους τομείς. Ε, λειτουργούμε σε προληπτικό και διορθωτικό επίπεδο ταυτόχρονα. Κρατικές μεταρρυθμίσεις ε, διαχείριση δημοσίων οικονομικών, ε, συνεργασία με οργανισμούς ε, καταπολέμηση διαφθοράς όπου είπε υπηρεσία εξωτερική δράση, έλεγχος από πλευρά του Κοινοβουλίου για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ταυτόχρονα και θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντεπλεσί, είναι σωστό από την επιβολή του νόμου, από την προοπτική της οργανωμένης εγκληματικότητας να κατευθυνθούμε προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι εγώ ήμουν στις αστυνομικές δυνάμεις και έχω περάσει πλέον στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διάφοροι φορείς ε, συμμετέχουν, ε, ε, η, τα ΜΜΕ, η ερευνητική δημοσιογραφία, οι κατακέλλοντες, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Υποστηρίζουμε με μια, ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπων. Θα ήθελα κλείνοντας να ε, πω ότι τρία πολύ επιτυχημένα παραδείγματα συζητήθηκαν σήμερα. Εγώ τεμάλα γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση, διότι ε, χρηματοδότησε σε πολύ μεγάλο βαθμό προς υποστήριξη αυτές τις πρωτόβουλες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα τροποποιήθηκε και ε, προσαρμόστηκε και εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες Λατινικής Αμερικής. Σημαντικό είναι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε δύσκολες περιπτώσεις Ουκρανία, Αζερβαϊτζάν. Όπως είπε και ο εισηγητής, θα πρέπει να καταμετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των μέσων μας. Να μην α, στεκόμαστε μόνο στα θετικά παραδείγματα όπως αυτά της Γουατεμάλας, αλλά να σταθούμε και στα πιο δύσκολες, στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, όπως είδαμε σήμερα. Ε, Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα και πάλι το λόγο για να ολοκληρώσουμε στον εισηγητή μας, τον κύριο Στρεβίτσιος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους, όλα τα μέλη του πάνελ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι παρουσιάσεις τους ε, και πραγματεύτηκαν πολύ διαφορετικές διαστάσεις του φαινομένου της διαφθοράς. Όταν μιλάμε για τις τρίτες χώρες, δεν μπορούμε να ε, ε, κλείνουμε τα μάτια και να ε, μην βλέπουμε τι συμβαίνει στις δικές μας χώρες, να εθελοτυφλούμε. Δείτε τα χρήματα της προσόδους από τη διαφθορά σε τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει σε δικές μας χώρες, γιατί αυτά τα χρήματα επενδύονται ε, στα κίνητα ε, ή στο χρηματιστήριο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, σε είδη πολυτελείας, σε πάρα πολλές χώρες, σε εταιρείε ανά τον κόσμο. αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την κοινότητα, την ένωση αξιών που έχουμε συγκροτήσει, θα πρέπει να ασπίσουμε και μία ένωση κατά της διαφθοράς. Να αναλάβουμε μελητή δράση, να ακολουθήσουμε καλά παραδείγματα για να ε, αναχαιτήσουμε τη ροή ε, παρανόμων προσόδων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εγκρίνει ε, ένα κώδικα καλών πρακτικών για να ελέγχει όλες τις επενδύσεις, όλες τις ροές, ε, οικονομικές ροές προς τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες και ελπίζουμε και προς τις τράπεζες του ΕΟΧ που προέρχονται από κρατικούς αξιωματούχους κρατικοί εξωματούχοι κάνουν πάρα πολλέ τέτοιε επενδύσει με βρώμικα χρήματα. Εάν εφαρμοστεί μια τέτοια πρακτική και γίνει τυπικό επίσημο έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουμε το καλό παράδειγμα τώρα. Κηρύττουμε, συντάσσουμε εκθέσει, αλλά ε, μπορεί σε κάποια κράτη να υπάρχουν καλά παραδείγματα. Ε, πρόσφατα νομοθεσία στο, στη Μεγάλη Βρετανία. Όμω, είναι μεμονωμένα τα παραδείγματα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση σε μεγαλύτερη κλίμακα, τίποτα δεν έχουμε να δείξουμε. Αυτό θα ήταν ένα δίχτυ ασφαλείας ε, κατά ε, τον, ε, του βρώμικου χρήματος. Απευθύνομαι στα μέλη του πάνελ. Σε πολλές χώρες η διαφθορά έχει γίνει και όργανο της πολιτικής. Οι ε, υψηλοί κρατικοί αξιωματούχοι ε, έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν διεφθαρμένοι για να, ε, για να είναι εγγυημένη η πίστη τους προς το, την κυβέρνηση. Στο περίπου. Δηλαδή, και όταν εμείς ε, συζητούμε με αυτές τις κυβερνήσεις και, τους, ε, και ε, βάζουμε το δάχτυλο επί του τύπου των ήλων και τους ρωτάμε τι κάνετε για να καταπολεμήσετε το φαινόμενο, εσείς μας λένε how about you, εσείς τι κάνετε, εσείς δέχεστε τα χρήματά μας στη συνέχεια σε επενδύσεις, σε αγορές, στα ακίνητα. Ε, αυτό μας απαντούν λοιπόν τα πράγματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους. Δεν πρέπει να είμαστε ε, ειλικρινής. Υπάρχουν χώρες που υποφέρουν από τη διαφθορά και τις ε, ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε για να δείξουμε το καλό παράδειγμα και να δώσουμε με για να ε, λύθουν σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Πριν ξαναδώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για ένα λεπτό αν θέλουν να απαντήσουν, να ακούσουμε τον κύριο Ντεμερσμέκερ που ζήτησε επίσης το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες μας που έλαβα μέρος στη δημόσια ακρόαση και να ευχηθώ στον Πέτρα Σοστρεβίτσιους καλή τύχη και καλή επιτυχία με την έκθεσή του. Γιατί η διαφθορά είναι ο καρκίνος των κοινωνιών μας. Και συμφωνώ και με την κυρία Αναγκόμες. Άλλωστε αυτό ήταν το βασικό μήνυμα και της έκθεσης της ε, του 2013. Δεν μπορούμε εμείς να στυλιτεύουμε και να δακτυλοδεικνύουμε τρίτες χώρες όταν ε, ε, δεν έχουμε συγγυρίσει πρώτα το του οίκου μας, όταν επιτρέπουμε πρακτικές διαφθοράς και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εμφανή ο σχετισμός διαφθορά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύω ότι αν άλλο εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε τι ρόλο μπορούμε να διαδραματίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, βασικός ε, ε, δωρητής και μίζων χρηματοοικονομικός εταίρος θα πρέπει να δείξει το παράδειγμα, να δώσει το καλό παράδειγμα και να παρέχουμε χρηματοοικονομική βοήθεια μόνο σε χώρες που κάνουν χρηστή διαχείριση των κονδυλίων. Το Ελεκτικό Συνέδριο κατέληξε το 2013 στο συμπέρασμα ότι εμείς ως βασικός οικονομικός εταίρος της ε, Δημοκρατίας του Κονγκό θα πρέπει να επιβάλλουμε περισσότερους όρους στη χώρα αυτή προκειμένου να παρέχουμε την αναπτυξιακή μας βοήθεια. Επιπλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Έχουμε και κανονισμό για το εμπόριο των όπλων. Παρέχουμε οικονομική βοήθεια σε κάποιες χώρες και ως αντιστάθμισμα οι χώρες αυτές οφείλουν να τηρούν τους διεθνείς κανόνες. Το Πακιστάν για παράδειγμα, πολύ καλή περίπτωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα προβλήματα που έχουμε στο Πακιστάν και θα πρέπει να τηρηθούν τα συμφωνημένα θέντα οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και να υλοποιούνται από, όλες ε, τις, ε, από όλα τα συμβαλώμενα μέρη. Πολύ ενδιαφέρουσα η προτάση κυρίας Πέτερς. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να τις εφαρμόσουμε βέβαια εμπράκτος. Δεν κατάλαβα πώς μπορούμε να καταγγέλουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υιοθετώντας αυτή τη νέα προοπτική, το νέο πρίσμα της διαφθοράς. Και τι αντίκτυπο θα έχει μια τέτοια προσέγγιση στη δικαστική πρακτική. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις διεθνείς κατευθυντήρες γραμμές στη νέα αυτή προσέγγιση και να ζητήσουμε από την ειδικό εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ να αναλάβει δράση. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τους μηχανισμούς ε, του σεβασμού των ε, διεθνών κανόνων και ίσως να ενισχύσουμε αυτούς τους διεθνείς κανόνες που είναι αρκετά χαλαροί ή τουλάχιστον δεν εφαρμόζονται σωστά. Και ε, επίσης η Ουκρανία που είναι στην 103η θέση του δίκτυ της ε, διεθνούς διαφάνειας ε, που περιλαμβάνει 167 χώρες. Είναι σχεδόν ουραγός. Είχαμε την Πορτοκαλή Επανάσταση, αλλά δεν έφερε και θεαματικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς που είναι η βασική για της Ουκρανίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη θεωρία υπάρχουν καλά σημεία, αλλά στην πράξη ελάχιστα αλλάζουν. και από επαφές που έχω με Ουκρανούς πολίτες γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες σε νομοθετικό επίπεδο για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς, θεσπίζονται μάλιστα και νέοι φορείς και νέοι θεσμοί, αλλά όλα αυτά θα παραμείνουν νεκρό γράμμα αν δεν αλλάξει η νοοτροπία. Αν δεν αλλάξει η κουλτούρα της διαφθοράς, η νοοτροπία που τροφοδοτεί τη διαφθορά. Ε, εξακολουθούν να ε, ε, λιμένονται την κατάσταση οι λίγοι ολιγάρχες και να κινούν τα νήματα στο κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση, ακόμη και σε επίπεδο προεδρίας της Δημοκρατίας. Βλέπετε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμπλεκόταν στα έγγραφα του Παναμά. Θα πρέπει το σύστημα να αλλάξει ριζικά. Αν δεν γίνουν τέτοιες ρηξικέλευτες αλλαγές, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση, να επιλυθεί το πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη ε, δουλειά και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες στην, Ουκρανία. Και φυσικά και οι δημοσιογράφοι δεν θα πρέπει να μειώσουν τις προσπάθειές τους γιατί είναι πολύ χρήσιμες. Δεν ξέρω αν θέλετε το λόγο, καλεσμένοι μας, θα ήθελα να πω κάτι. Ένα λεπτό παρακαλώ καθένας, γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Παρακαλώ. Με την ίδια σειρά που λάβατε το λόγο πριν. Καλώς να απαντήσω στην ερώτηση του εισηγητού. Καταρχήν, διαφάνεια και απέτηση δημοσίευσης, αποκάλυψης. Αυτά είναι οι λέξη κλειδιά. Ε, και νομίζω ότι είναι το πιο, αναλογικό, ε, μετριοπαθέ και αποτελεσματικό μέσο. Αποκάλυψη των συναλλαγών. Τώρα με τι μορφές, ε, ε, νομικές μορφές θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο. Καταρχήν, μία απόφαση πλαίσιο για μέτρα ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων υπάταξης τη διαφθοράς. Επίσης, Εμπορικέ προτιμήσει ε, και τρίτον η Ευρωπαϊκή Ένωση ω περιφερειακή οργάνωση μπορεί να προσχωρήσει στην σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς και να συμπεριληφθεί η διαφθορά και στο σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνδυαστεί με τα σχέδια δράση που απαιτούνται με βάση τι αρχέ ράγκη των Ηνωμένων Εθνών για τι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Indeed, I can just Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε η προλαλή σα, Αρχές Ρέγγι δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών και έργο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Έχουμε ούριο άνεμο, πολύ περισσότερο σχέση με τον παρελθόν. Είχαμε, έχουμε και την παγκόσμια διάσκεψη κορυφή για την πάταξη Διαφθορά. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη φόρα που πήραμε, αυτή την όθηση που δημιουργήθηκε και είναι μοναδική και η ευκαιρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει αυτόν τον αγώνα. Και θα πρέπει να δράξει αυτή την ευκαιρία και να αποδείξει την στράτευσή τη υπέρ τη καταπολέμηση τη διαφθορά και εντό και εκτό αυτή. Και να υιοθετήσει πρακτικού μηχανισμού χρήσιμου, αλλά και να το συμπεριλαμβάνει στι διμερεί εμπορικέ συμφωνίε ή συμφωνίε χρηματοδότηση. Θα πρέπει ε, πρώτα να γίνει δεκτή η απέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετά να εφαρμοστεί πιο εκθετικά σε πιο λεπτομεριακούς μηχανισμούς. Ευχαριστώ. Э, большое спасибо Ευχαριστώ. Πολλά από αυτά που αναφέρατε είναι σωστά και στοιχειοδετημένα. Εγώ θα ήθελα να μείνω ε, σε τρία συγκεκριμένα σημεία ως προς την κατάσταση στην Ουκρανία. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ε, τα μέτρα που παίρνουμε θα πρέπει να στοχεύουν τους ανώτατους αξιωματούς παραβα... που παραβαίνουν τον νόμο και όχι ε, το γενικό κοινό. Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση και με την εξαίρεση ε, για την υποχρέωση θεώρηση. Εγώ έπρεπε να πάρω βίζα για να έρθω. Οι αθλητές, οι φοιτητές, οι μαθητές το ίδιο. Οι αξιωματούχοι όμως δεν χρειάζονται θεώρηση. Ε, όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς ε, μετακινούνται χωρίς θεώρηση. Έχουν τις πολλαπλές, τη θεώρηση πολλαπλής εισόδου του Σέγγεν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το σύστημα. Πρέπει να βοηθά το γενικό κοινό και όχι ε, να επιβραβεύει αυτούς τους αξιωματικούς όπως κάνει τώρα. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά το θέμα των κυρώσεων για την Ουκρανία, για την Αιγύπτο, ε, για κυβερνήσεις που έχουν ανατραπεί. Εξ πώς συζητεί το θέμα μετά από τις επαναστάσεις. Γιατί κανένας δεν σχολιάζει, σχολιάζει αυτό το ζήτημα όταν ήταν ακόμη στην εξουσία αυτοί οι άνθρωποι, είναι σημαντικό να γίνουν ρυθμίσεις ούτως ώστε οι ακτιβιστές και οι δημοσιογράφοι να μπορούν να, να μεταδίδουν τις πληροφορίες την ώρα που συμβαίνουν τα πράγματα. Όταν είναι στην εξουσία αυτή η άνθρωποι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό διότι ε, οι κυβερνήσεις ε, φροντίζουν να μην διαρρέουν τις επιβαφορίες. Και τρίτον, ε, τα, το βρώμικο χρήμα, ε, είπατε, δαπανάτε στην Ευρώπη. Στο Χάρκιβ, παραδείγματος χάρη, γιατί αναφέρθηκα στον Κέρνς στην παρουσίασή μου, έχει αγοράσει όλο τον Μπάντεν Μπάντεν στη Γερμανία. Και στο Χάρκοβο ε, πολλοί γνωρίζουν αυτή την κατάσταση τι λείπει λοιπόν μας λείπει ένα μέσο, ένα εργαλείο που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ούτω ώστε να τεκμηριωθούν αυτά για να μπορέσει να ε, ακολουθήσει και η δίωξη. Ακίνητα στο Λονδίνο ή ε, στην ε, Νότια Ισπανία ή στη Γαλλία πολλοί επενδύουν στον τομέα των ακινήτων. Χρειαζόμαστε τους ε, ε, καταγγέλλοντες, ε, τους ακτιβιστές και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν ένα μέσο για να μπορέσουν να μας μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτή την ανταπόκριση περιμένουμε από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και να σα πω ότι σε σχέση με τι ερωτήσει του εισηγητή έχω πολύ συγκεκριμένη πρόταση για το Αζερβαϊτζάν. Η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή πολιτική και οι εθνικοί και οι ευρωπαίοι βουλευτέ θα πρέπει φυσικά να έχουν μια φυσικά σωστή συμπεριφορά σε σχέση με χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν. Εδώ είχαμε κάποια προβλήματα με βουλευτές ε, που ε, έκαναν επισκέψεις στο Αζερβαϊτζάν. Έξι ε, βουλευτές παραβίασαν τον κώδικα διοντολογίας κατά τη διάρκεια αποστολών στο Αζερβαϊτζάν, αλλά δεν, πειθαρχική δράση δεν αναλύθηκε εναντίον τους, οπότε είναι η διπλωματία χαβιάρη, έτσι την ονομάζουμε εμείς. Ε, αυτά, αυτές οι πρακτικές και εδώ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να σταματήσουν οποιαδήποτε ε, ταξίδι προς το Αζερβαϊτζάν που εμπλέκονται αξιωματούχοι ε, πρέπει να, είναι, να, υπάρχουν, να έχουν και δικλείδες ασφαλείας, ε, να είμαστε σίγουροι ότι είναι άμεμπτη η συμπεριφορά όλων των ε, βουλευτών. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Ε, μία μικρή παρέκβαση. Ε, ε, λέτε, Lux Leaks, ε, όλα αυτά τράβηξαν την προσοχή των ΜΜΕ. Όμως δεν είναι η το μοναδικό θέμα που δεν, δεν είναι τόσο σεξι, αλλά δεν έχουν τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ. Πέρσι οι, αυτούς που έχουμε εγκαταλείψει, αυτοί που έχουν ε, πέσει θύματα έξωσης. Ε, Παραδείγματο χάρη, η Παγκόσμια Τράπεζα βρήκε ότι 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει ε, το σπίτι τους, τα κτήματά τους και δεν μπορούν να ζήσουν, να βγάλουν τα προστοζήν πλέον. Απλώς θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες έρευνες πολύ σημαντικέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν ασχολείται κανείς με αυτές τις περιπτώσεις γιατί δεν είναι τόσο ελκυστικές. Μετά από αυτή την παρέκβαση θα ήθελα να σας πω πως με την ερευνητική δημοσιογραφία, όπως στην περίπτωση LuxLeaks και Panama Papers, Χωρί τον καταγγέλλοντα δεν γίνεται τίποτα. Εάν δεν μα δώσει τα έγγραφα, αν δεν υπάρχει αυτό ο θαραλέο που θα τα παίξει όλα, ό,τι έχει κερδίσει σε ολόκληρη τη ζωή για να μπορέσει να φέρει την αλλαγή στην κοινωνία, χωρί τον καταγγέλλοντα, δεν θα μπορούσαμε εμεί ε, να έχουμε μεγάλη επιτυχία. Καταλαβαίνω πως ε, είναι σημαντικό για το Κοινοβουλίο το όλο ζήτημα της οδηγίας για το απόρριτο. Μην ξεχνάτε όμως να προστατεύετε με το απόρριτο και τους ε, καταγγέλλοντες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Πώς το μέλλον θα τους προστατεύσει καλύτερα. Αν δω τους λίγους που ξέρουμε, τον Τελτούρ, Αντών Τελτούρ, από τα Λάξ τον Ιούνιο στο Λουξεμβούργο ότι το καταδικάστηκε. Ο κύριος Φαλτσάνη είναι στην Ελβετία, το ξέρουμε αυτό. Επίσης στη φυλακή. Κάποιοι που διέρευσαν ε, ε, ε διπλωματικές ειδήσεις στο Swiss Leaks ε, επίσης ε, είναι στη φυλακή και άλλοι αποφάσισαν, επειδή δεν θέλουν να είναι οι επόμενοι στη σειρά, να μην παραμείνουν ανώνυμοι μέχρι που να υπάρξει καλύτερη προστασία για τους καταγγέλλοντες, αποφασίζουν κάποιοι να μην ε, δώσουν τα έγγραφά τους στη δημοσιότητα. Λένε ότι εγώ προτίθεμαι να ανταδώσω δώσω στις κυβερνήσεις, αλλά παρακαλώ να φροντίσετε πρώτα απ' όλα να κατοχυρώσετε την προστασία των ε, καταγγελόντων. Και αυτό ήθελα εγώ να τονίσω, πόσο σημαντική είναι αυτή η πτυχή. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Μαροκίνα. Ε, αν ε, εξακολουθεί να μας παρακολουθεί από το Skype και υπάρχει σύνδεση μαζί του. Μπορείτε και εσείς να πείτε κάτι αν θέλετε κύριε Μαροκή. Sí, adelante. Sí, adelante, adelante. Estamos concluyendo. Puede usted, tiene usted un minuto para... Τελειώνουμε την ακρόαση. Παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Έχετε και εσείς ένα λεπτό. Τελικά σχόλια, αν με ακούτε. Να με όγε. Να με όγε. Με σκούτσα. Να. Δεν ακούει ο κύριος Μαροκίν. Buenas tardes, otra vez. No. Ni yo a él tampoco le escucho. Ούτε εκείνο μα ακούει, ούτε εμεί τον ακούμε. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο στη σύνδεση Skype. No, él está hablando, él está hablando. Ok. okay. Thank you. Bueno, pues eh, lo siento porque no, no, no les. Κρίμα, κρίμα, αλλά δεν έχουμε ήχο από τον κύριο Μαρόκιν. Πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε. Στείλτε του ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για να ξέρει ότι ολοκληρώσαμε. Και ο κύριος Αστρεβίτσιος πρέπει να τρέξει στο αεροδρόμιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τις έγκριτες τους παρουσιάσεις. Εμείς ε, είμαστε στρατευμένοι και θα συνεχίσουμε το έργο μας, οπότε σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ε, θερμά ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη Δημόσια Κρόαση. Bueno, vamos a ver si acabamos con el último punto. Ας προσπαθήσουμε τώρα να διεκπαιρεώσουμε και το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης μας. Την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, τα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Ετήσια έκθεση του 2015. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ, υπενθυμίζοντάς του ότι μία ε, συνάντηση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για διαβούλευση θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου, 4 με 5.30, ημέρα Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, στην αίθουσα ΑΣΠ 5G305. Φαντάζομαι θα έχουν ενημερωθεί οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τη συνάντηση αυτή με τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ και θα ήθελα να του δώσω το λόγο ευχαριστώντας τον εκ των προτέρων για το έργο που κάνει στην έκθεσή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να μου επιτρέψει να κάνω κάποιες αγωγικές παρατηρήσεις στην έκθεση και θα σας μιλήσω και για το τι μέλη γενέστε. Ε, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι μπορώ να εργαστώ εδώ, διότι μου αρέσει πολύ η συστηματική σκέψη του κυρίου Παντσιέρη και του κυρίου Πρέντα και οι δύο αποφάσισαν να συντάξουν μια συστηματική θα τη χαρακτήριζα έκθεση μια έκθεση με μέθοδο, με σύστημα ε, και το θέμα δεν είναι να μπούμε σε λεπτομέρειε, αλλά να ακολουθήσουμε περισσότερο μια συγκεκριμένη μέθοδο. Αυτό έγινε στο παρελθόν και εγώ πάνω σε αυτή τη γραμμή θέλω να συνεχίσω. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, τα εργαλεία τα οποία είναι καθοριστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε μια καλή αξιολόγηση. Υπάρχουν θέματα τα οποία έρχονται και επανέρχονται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα όπως, ε, παραδείγματο χάρη, τι σημασία έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για το εμπόριο, για τις επιχειρηματικές σχέσεις θέματα που άπτονται της αναπτυξιακής πολιτικής, των ανθρωπιών δικαιωμάτων, της θανατικής ποινή επίσης, αυτό πάλι μας απασχολεί ιδιαίτερα και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που δεν είναι καινούρια, τα οποία όμως ε, προβάλλονται περισσότερο. Πρόκειται κυρίως για το ρόλο που διαδραματίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περιπτώσεις και περιόδους κρίσης και συγκρούσεων. Ε, επίσης υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με τα εγκλήματα πολέμου, ο ρόλος του φερόμενου Ισλαμικού κράτους και ένα άλλο θέμα, ε, ανθρώπινα δικαιώματα και αντιτρομοκρατία. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Στην Υποεπιτροπή είχαμε μια σχετική συζήτηση ε, παραδείγματος χάρη σε σχέση με την χρήση των ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών και αυτά πάλι σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ ότι το θέμα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ πιο προσεκτικά. Γιατί τίθεται το ερώτημα ε, κατά πόσον όλα αυτά άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι κατοχυρωμένα ε, στα ε, συντάγματά μας. Αν θέλετε, λίγο πολύ, αυτό είναι το περιεχόμενο που θέλω να δώσω στην έκθεση. Έχω ήδη κάνει κάποιες ε, πρώτες σκέψεις, κάποια διατύπωση και... Θα σας υποβάλουμε την έκθεση την επόμενη εβδομάδα και κατόπιν στις 26 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί η έκθεση αυτή στην υποεπιτροπή μας. Προηγουμένως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, θα λάβει η χώρα η συνάντηση με τις ε, ΜΚΟ, όπου όλοι οι συνάδελφοι, αλλά κυρίως οι ηγητές είναι προσκεκλημένοι για να λάβουν μέρος. Όπως ήδη το είπε η Πρόεδρος, αλλά το επαναλαμβάνω και εγώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. 6 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η συνάντηση, ε, τρίτη απόγευμα. Ε, σας καλώ λοιπόν να έρθετε όλοι σας, γιατί τις ε, απόψεις που θα εκφραστούν, επιθυμώ εγώ να τις συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Μετά θα πρέπει να καθοριστεί η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα κατατεθούν οι σχετικές τροπολογίες και η συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στην Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου. Όλα αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να ψηφίσουμε στις 14 Νοεμβρίου και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα, βεβαίω αυτό εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε πριν από το τέλο του έτου να κατατεθεί η έκθεση και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Αυτά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ε, θα υπάρξουν βέβαια και συγκεκριμένε προσκλήσει για συναντήσει των σκιωδών. Ε, εισηγητών. Δεν έχουμε καταλήξει όμως ε, σε αυτά. Ε, για το Πέπε Ρόβολτ, για το Ίσιαρ ΧΕΝΚΕΛ, Άλντε, Σάκε, Πράσινη, Λοχπίλα, Γκούε. Δεν έχει ακόμα. Α, εσείς. Εντάξει, εσείς. Και Ιγνάσιο Κοράο για EFDD. Αυτά όσον αφορά στα οργανωτικής φύσεως θέματα, στη δομή του κειμένου και παρακαλώ να μου καταθέσετε προτάσεις, θέματα που είναι σημαντικά για σας, να μου τα αναφέρετε. Σας είπα και πάλι ότι πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο είναι να καθορίσουμε τη μέθοδο, το σύστημα, γιατί Αλλιώς μπορούμε να προσθέσουμε και άλλου είδους προτάσεις. Υπάρχουν τα κατεπήγοντα, υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στο να δώσουμε ε, σάρκα στο πλαίσιο αυτό. Ωραία, θα δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ε, όχι μόνο στους και ηγητές. Ε, ο κύριος Γκζιπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα αντικαθιστώ τη συνάδελφο Κριστ Τροβόλ, που είναι η σκιώδης ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ για αυτά που είπε ότι η δική του έκθεση είναι η συνέχεια των προηγούμενων ε, εκθέσεων των συναδέλφων Πρέντα και Παντσέρη. Δηλαδή δεν θα ε, βρίσκουμε τον τροχό με την τελευταία έκθεση, απλώς ε, συνεχίζουμε τη φυσική πορεία των προηγούμενων τάσεων που επισημάναμε στις προηγούμενες μας εκθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ καλό θετικό το σημάδι που δίνει ο εισηγητής Βάιντεν Χόλτσερ. Επίσης ε, και η επιμέρους παρατηρήσεις για το σε ποιους τομείς επικεντρωθεί ε, είναι πολύ θετική ονή για την μεταγενέστερη έγκριση της έκθεσης. Αυτές είναι οι προσωπικές μου απόψεις. Τώρα, η συνάδελφος Κρίς ε, Χαουτεροβόλ θεωρεί ότι το 2015 ήταν ε, μια δύσκολη χρονιά με πολλές προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με πολλά θέματα που άπτονται και του προσφυγικού, αλλά και με την εμφάνιση, την έξαρση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Και είδαμε επίσης ε, τις ε, διώξεις ε, και των μειονοτήτων κυρίως των θρησκευτικών. Με τις τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις έχουμε κατάφορες και σοβαρές καταστρατηγήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χαιρόμαστε για την έγκριση του νέου σχεδίου δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019. Επίσης, ε, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη της ανεξιθρησκείας και της ελευθερίας ε, θρησκευτικής ε, πίστης. Αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε στη σχέση με τις τρίτες χώρες, αλλά και στις πολυμερείς μας συναντήσεις. Επίσης, θα πρέπει στη συνεργασία μας να προωθούμε τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Με ικανοποίηση η κυρία Ροβόλ θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013 για το ίδιο θέμα αποτέλεσαν προτεραιότητα και του νέου σχεδίου από το 2015 και μετά. Και θα πρέπει να ε, συνεχιστούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και να εφαρμοστούν και στις επόμενες χρόνιες. Επίσης θα έχουμε την 70η ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εκεί το ψήφισμα για την αλεξιθρησκεία και την ε, ελευθερία πίστης με πρόταση Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε δεκτό ε, με συνένεση στη Γενική Συνέλευση, την 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, το θέμα, γιατί δεν είναι εύκολη αποδοχή με συνένεση οποιασδήποτε πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, το 2015 είχαμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνευ προηγουμένου άφηξη μεταναστών και κυρίως προσφύγων. Και θα πρέπει να τονίζουμε και πάλι και να διετρανώνουμε την προτεραιότητα που δίνουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε με θέσπιση μηχανισμών όπως το Ταμείο για την Αφρική το Trust Fund για τη Συρία, το Καταπίστημα για τη Συρία, αλλά και η συμφωνία με την Τουρκία για τη βοήθεια των σύρων προσφύγων εκεί. Επίσης, ε, κάποιες ε, ενέργειες που γίνονται στη θάλασσα, σωστικές ενέργειες που το 2015 μας επέτρεψαν να διασώσουμε πάνω από 7.000 ε, ανθρώπους. Βέβαια, οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι ε, ο μεγάλος αριθμός των διασωθέντων στις ε, όχθες της Λιβύης δείχνουν ότι είναι πολύ ήταν πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των θυμάτων των λαθροδιακίνητων προσφύγων. Και δυστυχώς αυτό το φαινόμενο εξακολουθεί να υπάρχει. Το ε, Νοέμβριο του 2015 το Συμβούλιο κατέληξε συμπεράσματα για την στήριξη της δικαιοσύνης διεθνώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρωτοστατεί στις διεθνείς πρωτοβουλίες ε, για την διεθνή διάσταση της δικαιοσύνης και μάλιστα με κυρωτικά κονδύλια χρηματοδοτούμε μεταξύ άλλων ε, σχέδιο αναπτυξιακό στο Κονγκό και επίσης το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη στήριξη που προσφέρουμε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μάλιστα το 2015 έχω, για το 2015 είχαμε αφιερώσει μια συνεδρίαση μας στο θέμα της συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε ό,τι αφορά το, τη δημοκρατία και τις εκλογές. Η κυρία Ροβόλ θεωρεί ότι είναι μία από, ένας από τους πυλώνες της Σωστή εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελεύθερε ανώθευτε εκλογές είναι απαραίτητη προϋπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τέτοιε διαδικασίες. Γιατί μόνο με ελεύθερες εκλογές μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα ένα κράτος με τους εσωτερικού του θεσμού. Και μόνο έτσι μπορούν να εφαρμόζονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σήμερα ε, στη δημόσια κρόση που είχαμε για το σχετισμό διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είδαμε και από αυτή την πτυχή το θέμα. Θα πρέπει να εξακολουθούμε να στέλνουμε αποστολές παρατήρηση εκλογών ως ε, σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, η κυρία Ροβόλ επισημαίνει την δέσμευσή της και την προσήλωσή της στο θέμα και την υπόσχεσή της για στενή και επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή με παρουσία της ε, σε όλες τις ε, συναντήσεις και σκέψεις εργασίας που θα γίνει για την περαιτέρω επεξεργασία της ετήσιας έκθεσης για το 2015. Σας ευχαριστούμε κύριε Ξύπ. Ο λόγος τώρα στην κυρία Βεριζιά εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Oui, merci. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας ε, που αν κατάλαβα καλά ακολουθεί τη γραμμή των Παντσέρη και Πρέντα των προηγούμενων εισήγητων και εγώ υποστηρίζω την ε, προσέγγιση να ξεφύγουμε αυτή τη λογική του καταλόγου και να επικεντρώσουμε τις προτάσεις μας σε συγκεκριμένους τομείς και θέματα. Τι με απασχολεί το ότι κατά τη γνώμη μου χρήσιμη είναι η έκθεση μόνο για να αυτοσυγχαρούμε για όλα τα καλά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως καλό είναι να τονίσουμε και που ακόμη υπάρχουν προβλήματα ούτως ώστε ε, να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προοδεύσουν στον τομέα των οποίων δικαιωμάτων. Ομολογουμένως έχω κάποιες ανησυχίες, ε, διότι βλέπω την Ένωση αλλά κυρίως και τα κράτη-μέλη της ε, να διαπραγματεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις για τις πωλήσει όπλων για τα μη επανδρομένα με κράτη που κατάφορα και προφανώς παραβιάζουν όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο πολέμου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας Ε, ναι, στο θέμα της τρομοκρατίας, στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, για να είμαστε σε εγρήγορση. Χρειάζεται ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, όμως ε, δεν μπορεί να δικαιολογήσει μαζικές παρεμβίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως ε, σε κάποιες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί σχέσεις ε, και τα κράτη-μέλη της ακόμη περισσότερο. Αυτές οι χώρες ε, πατάσουν κάθε ε, αντίθετη γνώμη, κάθε προσπάθεια εκδημοκρατισμού. Μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα είναι το επόμενο θέμα. Αυτή την έκθεση που πρέπει να την εγκρίνουμε το Σεπτέμβριο είναι, είναι νομίζω σημαντικό να ε, τονίσουμε ότι η ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βοηθήσει αυτές τις χώρες που αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές δροές να αποκτήσουν ένα οπλοστάσιο που θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν το πρόβλημα. Έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Δεν ήθελα σαν τον Πρεβέρ να κάνω ένα κατάλογο δικαιώματα γυναικών, ε, ελευθερία ε, έκφραση απόψεων, δικαιώματα ΛΟΑΔΜ. Βλέπω την κατάσταση ε, με τα δικαιώματα των γυναικών στην Λατινική Αμερική. Είναι λίγα ανησυχητικέ καταστάσεις που βιώνουν οι γυναίκες εκεί και μήπως θα έπρεπε να στρέψουμε το πλέον μας και σε άλλες υπήρους, υπήρους που έχουμε πολύ καλές σχέσεις, για να τους βοηθήσουμε να προοδεύσουν σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρέντα. Δεν ζητήσατε το λόγο. Ναι, ναι. Νόμιζα ότι προηγούνται οι συνάδελφοι από τι άλλε Δεν είναι κανένας εδώ. Εγώ τρία πράγματα πολύ απλά θέλω να πω. Πρώτον, Κύριε Χόλσερ, ε, ε, σας συγχαίρω για την πρόθεσή σας ε, μέχρι το πέρας του τρέχοντος να καταφέρουμε να ψηφίσουμε. Είναι και αυτονόητο. Πριν το τέλος του 16 να ψηφίσουμε την έκθεση για το 15. Λοιπόν, ελπίζω ότι αυτά που συνέβησαν στο 2015 θα αναφερθούν χωρίς να είναι επιμολυσμένα από τις εξελίξεις του 2016. Επικαιροποιούμε βερβολικά ορισμένες φορές τον πολιτικό μας λόγο μια κατάσταση που όμως περιγράφει τα δεδομένα του 2015, έχει περάσει ένας χρόνος. Είναι ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος να μην είμαστε ακριβείς. Δεύτερον, ε, βάσει και της παρελθούσας μου εμπειρίας, ξεπλάγει, ε, όταν διαπίστωσα πως ε, οι αγαπητοί συνάδελφοι από την ΤΕΒΕ και τη ΦΑΜ λίγες ώρες πριν την ψηφοφορία υπέβαλαν γνωμοδοτήσεις που υπερβαίνουν και την έκθεσή μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε. Εάν μας απασχολεί λοιπόν πραγματικά ε, η κατάσταση με τα δικαιώματα των γυναικών και όντως είναι ανησυχητική, μήπως να αφήσουμε και την Επιτροπή Γυναικών να γνωμοδοτήσει εγκαίρως. Ε, τι κάνουμε εμείς ε, πολύ καιρό ασχολούμαστε με το ζήτημα, αφιερώνουμε ε, μία-δύο παραγράφου ε, σε αυτό το ζήτημα και έρχεται η Επιτροπή Γυναικών με 45 παραγράφου για τα δικαιώματα των γυναικών. Θα το δώσουμε σε κάποιον και θα, θα αναρωτηθεί ποιο κάνει τι εδώ πέρα. Ποιο ε, ε, είναι καθήλυν αρμόδιο. Τώρα λέω τον πόνο μου γιατί θέλω να ρυθμιστούν ε, αυτά τα προβλήματα. Τα λέγαμε και στο παρελθόν, δεν διορθώθηκε η κατάσταση. Τελικά δεν ε, μπορεί να κάνει το διαβάσει κανένα στο έγγραφο. Καν, ποτέ, κανένα δεν συνάντησα που να μου είπε χάρηκα, πραγματικά το χάρηκα που διάβασα την έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όλοι είναι, πώς να το πω, όχι πολύ θετικοί ε, στις... Ε, εκτιμήσεις τους. Ε, δεν πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Τι τους δίνουμε να διαβάσουν. Για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να είναι εύληπτο, ευανάγνωστο και να εκλαμβάνεται ως χρήσιμο το κείμενο από τους ε, αναγνώστες. Τρίτον, προσπάθησα και πέρσι να τα πω και να επιμείνω. Ευχαριστώ τις πολιτικές ομάδες περιπτώντος γιατί με στήριξαν. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να τονίσουμε το ζήτημα του κράτους δικαίου, των κανόνα του κράτους δικαίου της δημοκρατίας σε ιδιαίτερα προβληματικά πολιτεύματα από πλευράς ε, δικαίου. Ε, και ως προς τους μετανάστες που δεν προέρχονται από δημοκρατικά πολιτεύματα. Δεν έχουμε τέτοιους μετανάστες. Να απαντάτε το φαινόμενο. Αν δεν υπάρχει πόλεμος, είναι πολιταρχικό το καθεστώς ε, ε, ή και χειρότερα, είναι δικτατορίες. Δεν έρχονται από αλλού οι μετανάστες τώρα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε. Μακροχρόνια παρέμβαση για να βοηθήσουμε αυτές τις κοινωνίες να αναπτυχθούν. Λοιπόν, από πολιτική σκοπιάς πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε όσες κυβερνήσεις έχουν κολλάσιμη δράση ε, να μεταρρυθμιστούν ώστε να ενισχυθεί ε, ο δημοκρατικός χαρακτήρας αυτών των ε, καθεστώτων. Δεν έχουμε φυσικά τη φιλοδοξία εδώ σε πολιτικό επίπεδο να ρυθμίσουμε προβλήματα πολύ βαθύτερα. Το πολιτικό ρόλο της ε, θρησκείας, παραδείγματος χάρη, ε, το, τις μαζικές μεταναστευτικές δροές. Δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε να τα λύσουμε εδώ τα προβλήματα. Το ευκολότερο είναι από πλευρά εκδημοκρατισμού των καθεστώτων να αποφασίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και μέσα από τις αποστολές παρατήρησης εκλογών τι μπορούμε να κάνουμε. Φερρυπίν. Κάθε χρόνο ε, έχουμε μια σημαντική υποστήριξη προς αυτές τις χώρες. Ε, παίρνει αυτή τη μορφή. Λοιπόν, ε, εδώ στην υποεπιτροπή μας θα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτά τα καθεστώτα από πλευρά εκδημοκρατισμού, παγίωσης της δημοκρατία, ε, παγίωση ε, του ε, νεότευκτου σε ορισμένες περιπτώσεις κράτους δικαίου, τι μπορούμε να κάνουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αυτοεπικρατικοί και τονίζουμε τα λάθη μας. Ε, μην ξεχνάμε κιόλα το χάσμα, το πελώριο χάσμα. Ε, μιλάμε για το κράτος ε, δικαίου, για το σεβασμό των ε, δικαιωμάτων. Ε, καταλαβαίνετε όμως για τους άλλους δεν είναι αυτονόητο. Δεν μπορούμε να εφεύρουμε εταίρου εκεί που δεν υπάρχουν. να τους βοηθήσουμε όμως μπορούμε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Τελικά ο κύριος Δερσμέκερ, παρόλο που δεν είχε ζητήσει αρχικά το λόγο, θα μιλήσει εκ μέρους της ομάδας του. Σας ευχαριστώ. Εν συντομία, ο κύριος Χέγκελ είναι ο σκιώδης ηγητής ε, της ομάδας μεταρρυθμιστών συντηρητικών από πέρσι γιατί θέλουμε να διασφανίσουμε μια συνέχεια. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω δυστυχώς ε, δεν βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Και αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα και αυτό είναι κάτι λίγο φαϊνότερο. Οπότε θα πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και επαγρύπνηση, να δούμε τις προτεραιότητές μας. Οι περισσότερες προέρχονται από τα θεμελιώδη προβλήματα που επισήμανε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εμείς ε, δίνουμε έμφαση στη νότια και ανατολική γειτονία, την κατάσταση στη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, την περιοχή του Καυκάσου, τη Νότια Ασία και θέματα που μας απασχολούν ιδιαίτερως, ελευθεροτυπία, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα δικαιώματα των παιδιών και είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Χέγκελ θα συνεχίσει το καλό έργο που ξεκίνησε από πέρσι και θα συμβάλλει επικοδομητικά στη διαμόρφωση της έκθεσης του κ. Βάιντερ Χόλτσερ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ο κ. Σέρι από την ΕΕ θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εν συντομία, θα ήθελα να πω ότι Άκουσα την ε, παρουσίαση που μας έκανε και ο εισηγητής ε, και τα σχόλια των μελών της Επιτροπής και θα, ακολουθήσουμε την διαδικασία που συμφωνήσαμε και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω από θεσμική άποψη σε αυτή τη διαδικασία, με τιμά ιδιαίτερως αυτό και χαίρομαι που η έκθεση θα λάβει υπόψη και τις προηγούμενες εκθέσεις και θα αποτελέσει τη φυσική συνέχειά τους. Και χαίρομαι που και οι δύο προηγούμενοι συγκητές Παντσέλη και Πρέντα ήταν παρόντες στη συζήτηση. Είμαστε και εμείς έτοιμοι και πρόθυμοι για επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Του τελευταίντος υπάρχουν και πολλά σημεία που θα αναλυθούν περαιτέρω στις ομάδες και με τα οποία συμφωνούμε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σίγουρα δεν βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο και σίγουρα δεν βελτιώθηκε το 2015. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα και της δικής μας έκθεσης, που όπως ξέρετε ήδη συζητήθηκε τον Ιούλιο. Και να πω ενημερωτικά δύο λόγια για την έκθεση. Ήδη το θεματικό τμήμα είχε εγκριθεί τον Ιούλιο και αυτό που είπε ο κύριος Πρέντα, το πόσο ευανάγνωστη είναι η έκθεση, αυτό πραγματικά α, ε, μας μιλάει. Γιατί συζητήθηκε στην Ολομέλεια και κάναμε ε, σημαντικές προσπάθειες ώστε η τελευταία μας έκθεση να είναι πιο ευανάγνωστη, πιο εμβριθής ε, και πιο συστηματική στον τρόπο που αναλύει τα πράγματα. Και είμαι υπερήφανος που για πρώτη φορά σε σχέση με τις προσπάθειες της τελευταίας πενταετίας θα έχουμε όσον νούπο και τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης με τη μορφή φυλαδίου. Και είναι πολύ σημαντικό και θα συμβάλλει στο να γίνει πιο ευανάγνωστη και να προβληθεί καλύτερα η δράση μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, για το γεωγραφικό τμήμα της έκθεσης, όπως ξέρετε η ετήσια έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, διαιρείται σε δύο τμήματα και το γεωγραφικό τμήμα δεν έχει εγκριθεί ακόμη, μόνο το θεματικό τμήμα εγκρίθηκε, αλλά και το γεωγραφικό τμήμα θα εγκριθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Τότε θα λάβετε και το γεωγραφικό τμήμα. Λόγω διαστάσεων μεγέθους, αλλά και για άλλους λόγους, δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, ούτε θα παρουσιαστεί ως φυλάδιο θα υποβληθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση. Αυτά ευχαριστώ θερμά και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία και περαιτέρω επαφές αν Ευχαριστώ κύριε Βάιτε Χόλτσερ. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ επικοδομητική συζήτηση. Δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία των διαφόρων τοποθετήσεων. Εγώ νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά που είπατε ε, θα τα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Βεβαίως ε, δεν μπορούσα να τα καταγράψω όλα ακριβώς. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε, όπως το έδειξε και ο συνάρφος κύριος ε, Πρέντα, γιατί κατ' ουσίαν εδώ δουλεύουμε και ως ιστορική Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο πρέπει να πάμε πίσω σε μια εποχή όπου δεν είναι δύσκολο να υπάρχει σαφής διαχωρισμός αλλά και ιστορικοί μπορούν να πέσουν στην παγίδα να ε, ε, αναλύουν την ιστορία με τρέχουσες και πίκερες απόψεις. Εγώ λοιπόν ε, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να πλατιάσουμε, θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πιο σαφείς και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να κοκορευόμαστε και να κομπορημονούμε, να προσπαθήσουμε λιγάκι να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία, τα χαρώ πολύ αν ε, ε, έρθετε να με βρείτε να συζητήσουμε αν έρχεστε τακτικά στις συναντήσεις των σκιωδών και επειδή το χρονοδιάγραμμα όπως σας είπα είναι αρκετά σφιχτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω τις τροπολογίες σας ή δυνατόν να τις καταθέσετε στα αγγλικά γιατί ε, στην περίπτωση αυτή θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε λιγάκι τη διαδικασία. Θα το ξαναπώ αυτό όταν θα φτάσει η στιγμή κατάθεση των τροπολογιών. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα και το ανέφερε ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ, αλλά να τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχήν, προπαρασκευαστική συνεδρίαση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, 6 Σεπτεμβρίου. Πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης ε, της Υποεπιτροπής θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών Λίγη στις 28 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Η εξέταση των τροπολογιών στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΑΦΕΤ Εξωτερικών Υποθέσεων, αν τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου, ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Και να πω κάτι στον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ. Το ανέφερε και ο κύριος Πρέντα. Μιλάμε για το 2015, να μην το ξεχνούμε. Και όταν μετά από 50 ή 100 χρόνια κάποιος ανατρέξει τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα χρειαστεί να το διαβάσει όσο και βαρετό και αν είναι οι ερευνητέ, θα πρέπει να καταλάβει ο ερευνητή ότι το 2015 ήταν η χρονιά που η Ευρωπαϊκή Ένωση Ίσως όχι η κοινωνία της, αλλά τα θεσμικά όργανα παλινδρόμησαν, έκαναν ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον τρόπο διαχείριση του θέματος και το πώς διαχειρίστηκε το προσφυγικό. Θα πρέπει να επισημάνω αυτό το σημείο καμπής που έγινε το 2015 και έγινε κάτι που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Ήταν πρωτοφανέ, γιατί πρόσφυγες είχαμε πάντα, αλλά δεν έφτασαν τόσο μαζικά στι ε, ακτέ μα. Αλλά ο τρόπο που διαχειριστήκαμε το προσφυγικό ήταν πραγματικά παλινοδία σε σχέση με την προάσπιση των αξιών μας. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο ιστορικός ερευνητής που μετά από χρόνια θα διαβάσει τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά, τελειώσαμε και καλό σας βράδυ. Σας. Looking forward, yeah? But not in English